Can Μήπως μπορούμε να αρχίσουμε οπότε και να καθίσετε ώστε να αρχίσουμε. Ακόμη έρχεται κόσμος βλέπω. Θα περιμένω 20 δευτερόλεπτα. Και θα αρχίσουμε με το σημείο 1 πρώτα. Αν δεν υπάρχουν σχόλια για την ημερήσια διάταξη, τότε να την εγκρίνουμε. Μπορεί εντωμεταξύ η έκθεση του κυρίου Κυρίλοφ, το θέμα του κυρίου Κυρίλοφ, να αλλάξει η θέση. Ίσως να πάει μισή ώρα ή νωρίτερα ή αργότερα. Γι' αυτό παρακαλώ να το ξέρετε ότι μπορεί να γίνει. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης, των προηγούμενων συνεδριάσεων. Εάν μέχρι το τέλος της σημερινής δεν ακουστούν σχόλια ή διαμαρτυρίες θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Τρία. Οι ανακοινώσεις της Προέδρου θα γίνουν αύριο μετά τη συνεδρίαση των συντονιστών και συντονιστριών. Και θα περάσουμε τώρα στο 4. Ανταλλαγή απόψεων με βάση ένα άτυπο έγγραφο που δημοσιεύτηκε στο οποίο, ε, το οποίο επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον, τη μελλοντική επανεξέταση του προϋπολογισμού και ιδιαίτερα το τμήμα του που αφορά την πολιτική συνοχής. Όπως είχα πει και γραπτός, όταν διέρευσε το έγγραφο αυτό, είχα ανακοινώσει και εξ ονόματός σας προς τον πρόεδρο της Επιτροπής και μετά και του Κοινοβουλίου ότι η δημόσια συζήτηση για την πολιτική συνοχή είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Επίσης, ως πρόεδρος της Επιτροπής Περίφ Ρέτζι έλαβα και διάφορες επιστολές από ενδιαφερομένους για την πολιτική αυτή, ιδιαίτερα συλλόγους και ενώσεις περιφερειών Γι' αυτό πρέπει να το ξέρετε, υπάρχει, υπάρχουν αντιδράσεις από πολλά όργανα και οργανισμούς σε ολόκληρη την Ένωση και δεν νομίζω ότι πρέπει σήμερα να συζητήσουμε το θέμα αυτό επί της ουσίας αν βέβαια μερικοί θέλουν να το κάνουν μπορούν έχουμε χρόνο για αυτό το θέμα μέχρι τις 4 αλλά βασικά πρέπει να εγκρίνουμε πώς, τι θα κάνουμε στο μέλλον, πώς θα αντιδράσουμε ως προς το έγγραφο αυτό που αντικατοπτρίζει τις απόψεις ορισμένων υπηρεσιών της Κομισιόν. Ακόμη κι αν αργότερα τροποποιηθούν, θα συζητηθούν πάντως και πρέπει και εμείς να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε ως αντίδραση στις απόψεις αυτές που νομίζω ότι δεν ανταποκρίνονται στις πεπιθήσεις της Επιτροπής μας ως προς την πολιτική συνοχής. Οι σχετικά νεότεροι συνάδελφοι στην Επιτροπή, καινούργοι, θα πρέπει να ξέρουν ότι έγινε μια ανάλυση της πολιτικής συνοχής μετά το 2013, τα τελευταία δύο χρόνια, η οποία ανάλυση και συζήτηση έγινε σε συνεννόηση με διάφορες κυβερνήσεις, ενδιαφερόμενους περιφέρειες, πόλεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έχουν οργανωθεί και υπουργικέ διασκέψεις για αυτό το θέμα, έχουν ληφθεί ορισμένες αποφάσεις Είμαστε λοιπόν στη μέση της συζήτησης του θέματος και όχι στην αρχή. Υπάρχουν δηλαδή εκπεφρασμένες απόψεις για την πολιτική αυτή. Και επειδή επίκειται η έγκριση, η θέση ενισχύει μάλλον της καινούργια συνθήκης που προσθέτει μία περιφερειακή διάσταση στην μαζί με την οικονομική και κοινωνική πρέπει να ταυτίσουμε ποιο νόημα θέλουμε να δώσουμε στη διάσταση αυτή και πώς θα συμπεριληφθεί, πώς θα ληφθεί υπόψη η περιφερειακή διάσταση. Επίσης η αρχή της επικουρικότητας θα ξεπερνάει πια, θα φτάνει και στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όχι μόνο το ευρωπαϊκό και το κρατικό. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μπουν στο παιχνίδι και νέοι παράγοντες. Όσοι δηλαδή είναι δραστήρια στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δεν μπορούν πια να αποκλείονται. Είναι και αυτοί πλέον τμήμα της νέας ευρωπαϊκής, του νέου ευρωπαϊκού τρόπου διακυβέρνησης ή governance όπως λέμε. Επίσης η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής θα έχει άλλη σημασία και βάρος πια, θα μπαίνει μέσα στο σύστημα της διαδικασίας συναπόφασης που θα είναι το κανονικό σύστημα απόφασης στο εξής. Αυτό σημαίνει όχι μόνο αυξημένο ρόλο του Κοινοβουλίου γενικότερα και ως προς την πολιτική συνοχής για την λήψη αποφάσεων και έγκριση των κανονισμών, αλλά θα δίνει και περισσότερο πολιτικό βάρος στο πολιτικό πρόγραμμα του Κοινοβουλίου. Και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να είμαστε πιο ενεργοί και στις συζητήσεις πριν την έγκριση του κάθε κανονισμού. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα της πολύ μεγαλύτερης σημασία που θα έχει στο εξής η πολιτική συνοχής και οι προτάσεις για μεταρρύθμισή της. Έχουν ακουστεί ιδέες, έχει διαρρεύσει και αυτό το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας της Κομισιόν, το οποίο δίνει μια άποψη για την πολιτική συνοχή που όπως σας είπα δεν συμφωνεί καθόλου με τις αρχές που οι περισσότεροι από εμά δέχονται και είναι βέβαια πολιτικός μη ορθών να αποκλείονται τα περιφερειακά και τοπικά επίπεδα αφού υπάρχουν εκεί παράγοντες ακαδημαϊκοί, επιχειρηματικοί, οργανώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας να μην αποκλειστούν αυτοί. Το έγγραφο αυτό είναι σαφές ότι αποκλείει από την πολιτική συνοχή στα επίπεδα αυτά και σταματάει στο κρατικό επίπεδο. Επίσης αποκλείει από την πολιτική συνοχή πολλούς στόχους που εμείς τους θεωρούσαμε πρωτεύοντες ως, ε, όπως η ανατομέα ανάπτυξη. Αυτά είναι πράγματα αλληλοσυνδεόμενα, δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε όπως κάνει το έγγραφο αυτό, ούτε καν για το θέμα των κλιματολογικών αλλαγών. Και φυσικά το ίδιο ανατομέα ανάλυση ισχύει και για τον προϋπολογισμό. Επίσης, στο έγγραφο αυτό βλέπουμε ότι αγνοούνται οι περιφερειακές ανισότητες γιατί αν μείνουμε στο εθνικό κρατικό επίπεδο τότε δεν μιλάμε πια για περιφερειακές ανισότητες ενώ εμείς τα τελευταία χρόνια το έχουμε ήδη, συζητήσει το θέμα των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών που σε πολλές χώρες είναι χτυπητές με την προσέγγιση λοιπόν της Κομισιόν αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη. Επίσης το έγγραφο δίνει τελείως άλλο βάρος στους πόρους που θέλουμε να διαθέσουμε. Το πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης μετακινείται σε μια διαχείριση κεντρικά από τις Βρυξέλλες Βλέπετε λοιπόν ότι με αυτά τα λίγα παραδείγματα του περιεχομένου του εγγράφου αυτού πιστεύω ότι κάτι δεν πάει καλά με την προσέγγιση του και γι' αυτό πρέπει να αντιδράσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να συμφωνήσουμε σήμερα με ποιον τρόπο θα αντιδράσουμε να αντιδράσουμε, επαναλαμβάνω, να είμαστε πιο ενεργοί, να παρουσιάσουμε το δικό μας όραμα για τον μελλοντικό προϋπολογισμό ως προς την πολιτική συνοχή ιδιαίτερα που μας ενδιαφέρει σήμερα και την περιφερειακή της διάσταση. Επίσης σκέφτηκα ότι ίσως το καλύτερο θα ήταν να υποβάλουμε προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν για ορισμένα από τα θέματα που ανέφερα όπως την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ή την πανενοσιακή κάλυψη της πολιτικής συνοχής γιατί ίσως δεν ξέχασα να πω ότι μία από τις σημαντικότερες πτυχές της πρώτης αυτής είναι ότι ο στόχος 2 εξαφανίζεται από την πολιτική συνοχή και ό,τι αφορά ακόμα και τις φτωχότερες περιφέρειες θα λύνεται κρατικά κατά αυτό το έγγραφο. Πρέπει και σε αυτό να αντιδράσουμε λοιπόν. Και μία δυνατότητα είναι ακριβώς η προφορική ερώτηση. Όχι αυστηρά για τον προϋπολογισμό ή για το κατά πόσον είναι επίσημο ή ανεπίσημο το έγγραφο αυτό, απλώς να αναφέρουμε δύο-τρία θέματα που θίγει όπως την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ίσως και μερικά άλλα, την κατανομή των πόρων γιατί επίσης περικόβει τα κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου στην πολιτική συνοχή. Τρία-τέσσερα θέματα δηλαδή να βάλουμε σε αυτή την προφορική ερώτηση και να ζητήσουμε στην Ολομέλεια συζήτηση. Αυτή είναι η πρότασή μου. Οι επιστολές που έστειλα θα σας πληροφορήσω αν έχουν λάβει απαντήσεως, αν λάβουν απαντήσεως, αν τύχουν απαντήσεως. Και έχετε τώρα το λόγο εσείς για να σχολιάσετε όποιος και όποια θέλει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να είναι πρώτο αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη διότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε ιδιαίτερα σοβαρά. Δεν ε, μας αφορά το θέμα ότι μιλάμε για ένα non-paper. Συνήθως αυτά τα άγγραφα έχουν μια κάποια επίδραση. Πρέπει να το εξετάσουμε, να δούμε αν μιλάμε για μια μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Έχουμε τις επιλογές ε, για το τι θα γίνει μετά το 2013. Να το δούμε λοιπόν επί της ουσίας. Εκείνο που είναι αξιοπρόσεκτο είναι το πότε παρουσιάζεται αυτό το έγγραφο. Διότι εδώ αλλάζουμε κατεύθυνση. Αυτό συνήθως γίνεται, δεν γίνεται στο τέλος μιας ε, θητείας, αλλά είναι και σημαντικό και επί της ουσίας. Αφενός έχουμε διάφορες ε, περιπλοκές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε τον παρόζο, τις απόψεις του, τις απόψεις των επιτρόπων και είναι σαφές, όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, ότι η περιφερειακή συνοχή θα αποτελέσει ένα απόσπαστο τμήμα της νέας συνθήκης. Ε, η ισπανική διερμηνία έχει κάποιο πρόβλημα. Μήπως τώρα διορθώθηκε. Ναι, α, εντάξει, συνεχίστε, συνεχίστε, ορίστε. Ευχαριστώ. Έλεγα λοιπόν ότι είναι πολύ περίεργο το χρονικό, η χρονική συγκυρία στην οποία παρουσιάζεται. Είναι πολύ σημαντικό να αντικατοπτρίζονται κάπου επί χάρτου αυτέ οι αλλαγέ. Και αυτό που είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε για το πώ θα ανταποκριθούμε σε αυτό και πώ ε, ανταποκριθήκατε και εσεί ω πρόεδρο στην ε, επιστολή σα, ε, νομίζω ότι οδεύουν προ τη σωστή κατεύθυνση. Αυτά που έχουν στο έγγραφο δεν συμφωνούν με αυτά που έχουν συμφωνηθεί στο παρελθόν και αυτά που εμείς ως Επιτροπή αλλά και ως Κοινοβούλιο εν γέννη θεωρούμε ότι είναι η σωστή άγουσα. Υπάρχει το θέμα της πολιτικής συνοχής, είναι μια έννοια την οποία αναπτύξαμε και εδώ για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συζητήσει και έχει καθορίσει σαφως το Κοινοβούλιο και δεν μπορεί κάποιο να έρθει εν μία νυχτή και να το αλλάξει. Και θα ήθελα μέσω ε, μόνο κυρία Πρόεδρε, να θέσω και μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να τους ρωτήσω λοιπόν να μας πούνε ακριβώς τι εννοούν με αυτό το έγγραφο. Διότι εμείς ε, τελικά από αυτό που διέρευσε στον τύπο μάθαμε τι λέει. Θα ήθελα λοιπόν η Κομισιόν να μας πει πού βρισκόμαστε, πού έχουμε φτάσει με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και αν ε, πρόκειται να εφαρμοστεί αυτό. Μιλάμε για ένα non-paper το οποίο εντάξει δεν θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσω, αλλά προ την ουσία σα ανέφερα ένα-δύο πράγματα, να αναφέρω και ένα-δύο πράγματα ακόμα. Για παράδειγμα, το μέλλον του στόχου 2, η ανταγωνιστικότητα. Αυτά τα χάνουμε από το έγγραφο εδώ. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν να υποβάλουμε μία προφορική ερώτηση για να τα θίξουμε αυτά τα θέματα και από εκεί και πέρα να έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας πει πώς σκοπεύει να τα συμπεριλάβει όλα αυτά. και να μην έρθουν με ένα εντελώ διαφορετικό έγγραφο μετά από δύο αργότερα. Η Επιτροπή Προπολογισμού βέβαια θα είναι αυτή η οποία θα καθορίσει ε, πού πληρούνται τα κριτήρια τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Ε, εγώ δεν νομίζω ότι πληρούνται τα κριτήρια. Το Κοινοβούλιο ε, πιστεύει εντελώ διαφορετικά πράγματα για αυτά τα πράγματα. Βέβαια, εγώ είμαι πλήρω μαζί σα στο θέμα τη επιστολή. Έχετε πλήρω την υποστήριξη και τη πολιτική μου ομάδα του ΕΛΚ για το θέμα και θα υποστηρίξουμε και την προφορική σα ερώτηση για την ουσία ουσία της πολιτικής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Όλμπριχτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να στηρίξω την προσπάθειά σας ε, για την επιστολή. Έχουμε βέβαια κάποιες αμφιβολίες, διότι το τελευταίο διάστημα βιώσαμε όλοι λίγο τις επιπτώσεις των επιστολών. Κάποιοι από εμά ε, θα θυμόμαστε ίσως την διάσημη επιστολή των 6 που δεν ήταν ένα επίσημο έγγραφο και αφορούσε όμως ε, πλήρως το θέμα του προπολογισμού. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω καταρχάς να γίνει αυτή η προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να απαντηθεί το θέμα στη διάρκεια της συζήτησης, αλλά εκ παραλλήλου νομίζω ότι είναι απαραίτητο να ετοιμάσουμε και εμείς τη δική μας τη θέση ανεξάρτητα από το τι πρέπει να γίνει βάσει της διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποτίθεται ότι είναι ενεργό εταίρο βάσει συνθήκη τη Λισαβόνα στη διαδικασία συναπόφαση. Επομένω, θα πρέπει να υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο θα ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα περιλαμβάνει κάποια σημεία για το τι πιστεύουμε εμεί για την πολιτική συνοχή. Δεν χρειάζεται λοιπόν να περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε και το Συμβούλιο εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάσει κάτι και το στείλει, για παράδειγμα, στην Επιτροπή των Περιφερειών, που ξέρουμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η νέα διαδικασία, αλλά εμείς να κάνουμε κάτι άλλο, να ετοιμάσουμε δύο σελίδες με τα σημεία τα οποία θεωρούμε ότι είναι υψή τη σημασία. χωρίς να λάβουμε υπόψη την επίσημη ε, κατάθεση του εγγράφου και να το ετοιμάσουμε ως θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να είμαστε δραστήριοι δηλαδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να σας πω ότι εγκρίνω απολύτως την αντίδρασή σας μετά την ανάγνωση αυτού του προσωρινού εγγράφου, του μυστηριώδους αυτού εγγράφου και νομίζω ότι έχετε επαναλαμβάνω απόλυτο δίκιο. Εγκρίνω επίσης τους όρους με τους οποίους απευθυνθήκατε στην Κομισιόν. Πράγματι, δεν είναι δυνατόν να μην αντιδράσουμε σε μια τόσο ριζική αλλαγή της πολιτικής συνοχής, ιδιαίτερα ως προς τις περιφέρειες. Πρέπει να αναλυφθούν πρωτοβουλίες. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ως το δυνατόν αποτελεσματικότερα και δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί η συζήτηση αυτή. Πάντως, έχετε την υποστήριξη της ομάδας Γκουε στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβετε και του συνόλου της Επιτροπής μας, ενώ έναντι της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Αλφόνση. Ναι, κυρία Πρόεδρε, και εγώ ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον προηγούμενο μιλητή. Στην ομάδα μας με ικανοποίηση βλέπουμε ότι φροντίσατε το θέμα και νομίζω ότι όσο το δυνατόν συντομότερα εκφράσουμε τις αντιρρήσεις μας τόσο το καλύτερο για να υπάρξουν και υπάρξει και συνέχεια διότι δεν αρκεί να πούμε κάτι πρέπει να ακουστεί και από τις περιφέρειες και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές που πρέπει να αντιταχθούν και αυτές σε αυτήν την τάση που θα καταλήξει τελικά σε διαδικασίες και δομές αναποτελεσματικές και που θα απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο από τον πολίτη. Εμείς είμαστε υπέρ αυτής της περιφερειακής διάστασης της πολιτικής συνοχής. Θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανισότητες των περιφερειών μέσα στα κράτη, πράγμα που είναι φανερό και στη Γαλλία και αλλού. Και επίσης θα θέλαμε τα περιφερειακά προγράμματα να μην εφαρμόζονται να μην εφαρμόζονται εις βάρος των ανατομέα προγραμμάτων αλλά παράλληλα. Επίσης είμαστε υπέρ αυτής της συνδιαχείρισης που είχε αρχίσει να διαφαίνεται από την προηγούμενη θητεία με τις περιφέρειες και νομίζω ότι μόνο σε αυτόν το, συνεχίζοντας σε αυτόν τον δρόμο θα μπορέσουν να λυθούν ορισμένα θεσμικά προβλήματα των πολιτών. Τέλος, Αν τελικά δημιουργούνταν μία προσωρινή επιτροπή για αυτό το θέμα, θα έπρεπε η επιτροπή μας να συμμετέχει πλήρως. Η κυρία Μανέσκου. Γαλλικά. Τι γαλλικά. Δεν το ακούω. Ε, ε, Κυρία Πρόεδρε, οποιαδήποτε αντίδραση θα εγκρίνεται θα μας βρει σύμφωνος διότι αυτό το άτυπο έγγραφο της ε, Κομισιόν δεν μας βρίσκει καθόλου σύμφωνος εφόσον περιέχει μέτρα που δεν θα βοηθήσουν καθόλου και τα νέα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δημοσιονομικά προβλήματα όπως ξέρετε πολύ καλά. Παραδείγματο χάρη η απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης κονδυλίων στήριξης και η μεταρρύθμιση των συστημάτων ελέγχου χρήσης των κονδυλίων αυτών. Αν το εξετάσουμε σε βάθος το έγγραφο αυτό θα διαπιστώσουμε ότι η Κομισιόν έχει μόνο μακροοικονομική και ανατομέα προσέγγιση και καθόλου μακροπεριφερειακή. Πράγμα το οποίο μας εκπλήσει διότι η συνθήκη της Λισαβόνας μιλάει ρητά για την περιφερειακή διάσταση και της δίνει πολύ σημαντική θέση. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος η πολιτική συνοχής να γίνει απλώς μία πολιτική φιλανθρωπίας και τίποτε παραπάνω. Ευχαριστούμε Τζον Μπάρτον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να συμφωνήσω με πολλά από όσα ακούσαμε σήμερα για την ε, άμεση αντίδρασή σας. Εγώ ως νέο μέλος πραγματικά ε, μένω κατάπληκτο από τον τρόπο που προχωράει το θέμα. Πολλοί άνθρωποι διαφωνούν για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι αυτό είναι ένα απτό παράδειγμα. Τα πράγματα πρέπει να είναι σαφή. Όταν παρουσιάζεται ένα έγγραφο, είτε υπάρχει διαρροή, είτε οτιδήποτε, πρέπει να ακολουθείται η σωστή διαδικασία. Νομίζω ότι η Επιτροπή μα έμεινε στο σκοτάδι, πλήρω στο σκοτάδι και αυτό είναι απαράδεκτο. Υπάρχουν ε, πολλές ε, ανησυχίες για την ε, χρηματοδότηση η οποία θα μπορούσε να σταματήσει εν μία νυχτή αν προχωρήσει αυτά τα όσα αναφέρει το έγγραφο και νομίζω ότι θα πρέπει να έρθει εδώ ο κύριος Μπαρόζο το συντομότερο δυνατό για να απαντήσει. Η επιστολή είναι καλή αλλά θα πρέπει να είμαστε λίγο σαφείς για το πού ακριβώς πηγαίνει η κατάσταση. Πολλοί μίλησαν, ακούσαμε πολλές ανησυχίες από όλο το Κοινοβούλιο για την αλλαγή κατεύθυνσης και νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε από το στόμα του ίδιου του κυρίου Μπαρόσο ότι ακριβώς ε, συμβαίνει. Θα πρέπει να έρθει είτε εδώ είτε αύριο αν γίνεται ε, ή το συντομότερο δυνατό για να ακούσουμε από αυτόν τι ακριβώς συμβαίνει. Ε, δεν είναι το θέμα της διαρροής, είναι θέματα τα οποία εξετάζονται. Θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς για το τι θα κάνουμε και εγώ ιδιαίτερα ανησυχώ για το πώς έχει κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μπράτπον. Σας ευχαριστώ. Και εγώ είμαι μέλος στην παρούσα επιτροπή. Αν και έχω κάπω το συνέστημα του déjà vu, γιατί και πριν από πέντε χρόνια που ήμουνα στην Επιτροπή Μεταφορών πάλι τα ίδια έβλεπα. Νομίζω ότι πάμε να καλύψουμε το ίδιο έδαφο που καλύψαμε προ όταν είχαμε συζητήσει τα τελευταία προγράμματα. Δεν έχω πρόβλημα με τα όσα λέχθηκαν σχετικά με το πώς προέκυψε το θέμα αυτό, πώς εμφανίστηκε το θέμα αυτό, αλλά υπάρχουν δύο ξεχωριστά θέματα εδώ. Το ένα είναι πώς μάθαμε περί της ε, αλλαγής κατεύθυνση της Κομισιόν, αλλά υπάρχει και το θέμα της ουσίας, περί της ίδιας δηλαδή της αλλαγής κατεύθυνση και αν όντω απηχεί την τρέχουσα νοοτροπία στην Επιτροπή, στην Κομισιόν δηλαδή, πάντως τότε πρέπει να συζητηθεί. Μιλώντας προσωπικά, και προερχόμενος από ένα κόμμα που είναι πολύ επιφυλακτικό σε ό,τι αφορά τα α, ωφέλη από αυτή την κυκλοφορία του χρήματος σε, στον τομέα αυτό, θα έλεγα ότι μάλλον σφραγίζει την καταδίκη οποιασδήποτε τέτοια πρόταση της Επιτροπής. Στην ουσία δηλαδή πάει να επανεθνικοποιήσει την πολιτική αυτή εάν όντω αυτό προτείνει η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν όντως απηχεί την νοοτροπία της αυτή τη στιγμή. Και τι γίνεται όμως στο ενδιάμεσο διάστημα, όταν βλέπουμε δηλαδή μια ουσιώδη πρόταση από τη στιγμή εκείνη μέχρι ότου να τη συζητήσουμε και πώς θα αποσπάσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με το ποιες ακριβώς είναι οι απόψεις της ίσως με την υποβολή προφορικής ερώτησης, με συζήτηση στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι αυτή η μέθοδος είναι πιο κατάλληλη. Πάντως, σε ό,τι αφορά το προς τα που κατευθυνόμαστε, για μένα είναι κάπως παράξενο ότι μια απερχόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε μια τέτοια ριζοσπαστική αλλαγή κατεύθυνσης. Η ερώτησή μου λοιπόν προς την Επιτροπή, προς την Κομισιόν δηλαδή, θα ήταν πρώτον από πού τα βρήκατε αυτά που βρέθηκαν δηλαδή, δεύτερον πού πηγαίνουν και τρίτο πότε και πώς το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να συζητήσει πλήρως ενήμερο τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ. Τώρα, τώρα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τίστε πρώτα το κοινοβουλιο θα μπορεσει να συζητησει πληρως ενημερο τα θεματα αυτα σας ευχαριστω τωρα τωρα ευχαριστω κυρια προεδρε κυριες και κυριοι συναδελφοι ειστε πρωτα το ερωτημα μήπως ίσως θα έπρεπε να είμαστε ικανοποιημένοι που βγήκε στην δημοσιότητα η πρόταση αυτή γιατί έτσι έχουμε και περισσότερο χρόνο για να την συζητήσουμε. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να συζητήσουμε την πρόταση αυτή. Το θεσμικό όργανο Κομισιόν έχει και καθήκον, εν πάση περιπτώσει, να κάθεται να σκέπτεται Πρόκειται τώρα για τι είδους έγγραφο. Πρόκειται για ένα μη έγγραφο, πρόκειται ίσως ε, για μια δοκιμαστική αν θέλετε ε, έκδοση της πρότασης αυτής για να δουν ποιες αντιδράσεις θα υπάρξουν. Πάντως υποστηρίζω κυρία Πρόεδρε την πορεία που προτείνεται. Με απασχολεί το ερώτημα εάν ίσως εδώ πάμε να κάνουμε τα πράγματα προθύστερα διότι εξάγονται συμπεράσματα χωρίς να προηγηθεί πρώτα μια λογική ανάλυση. Κανονικά πρέπει πρώτα να γίνει μια ανάλυση των ε, συνεπειών. Όπως για παράδειγμα και με την αντιπροσωπεία προς τη Μαδέρα που ε, πρότεινε ο κ. αυτά έχουν ε, αποβεί επιτυχή στο παρελθόν. Αλλά εδώ δεν έχουμε εμπειρίες στα, σε, σε σχέση με τα έργα αυτά. Δεν έχουν ακόμα δαπανηθεί καν τα κονδύλια. Πώς ε, λοιπόν τώρα θα κριθούν τα μέτρα αυτά για την περίοδο αυτή όταν ακόμη δεν έχει πραγματικά αρχίσει να εκτελείται. Νομίζω λοιπόν και εγώ ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια σε βάθος ανάλυση πάνω στην οποία να μπορέσουμε να βασίσουμε και οποιαδήποτε πολιτική για το μέλλον. Κύριε Μπρόν. Ε, ευχαριστώ. Δεν είμαι κι εγώ ε, σίγουρο σχετικά με το καθεστώς του εγγράφου αυτού, αλλά θα μου έκανε εντύπωση η Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού να έχει ε, εκδώσει τέτοιο έγγραφο χωρίς να έχει πρώτα συνεννοηθεί με τις άλλες Γενικές Διευθύνσεις της Κομισιόν. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σωστό να υπάρξει ταχεία αντίδραση εκ μέρους μας. Και καλά κάνατε και βάλατε και το θέμα σήμερα στην ημερησία διάταξη. Διότι πολλοί θα ανησυχήσουν από τις προτάσεις αυτές. Θα θυμάστε ότι προ ετών είχαμε ακούσει παρόμοιες προτάσεις από τις χώρες μέλη, με στόχο δηλαδή την επανεθνικοποίηση της ε, περιφερειακής πολιτικής. Την είχαμε τότε αποκρούσει την πρόταση αυτή και τώρα θα πρέπει να την αποκρούσουμε. Αλλά φαίνεται η Επιτροπή να υποβάλει πάλι παρόμοιες προτάσεις. Από την δική μου χώρα, την Ουαλία, γνωρίζω ότι πολλοί ανησυχούν και οι τέσσερις Ουαλοί βουλευτές του Κοινοβουλίου και ο Πρωθυπουργό μα και αναπληρωτής Πρωθυπουργό τη Ουαλία εξέφρασαν τι ανησυχίε του. Το μέγα λοιπόν θέμα για μένα είναι πώ αντιστεκόμαστε στις προτάσει αυτέ που περιέχονται στο έγγραφο. Και αυτό που νομίζω ότι χρειαζόμαστε είναι μια συντονισμένη προσέγγιση. Να συνεργαστούν και οι τοπικέ αρχέ των περιφερειών μα όσο μπορούν, ώστε οι ίδιε οι περιφέρειε να συνεργαστούν για να αντιδράσουν στις προτάσεις αυτές. Και βεβαίως η παρούσα Επιτροπή και οι Ευρωβουλευτές από τις ε, θυγόμενες περιφέρειες να συνεργαστούν όσο γίνεται στενότερα. Χρειάζεται κάποια συζήτηση λοιπόν για να δούμε ποιο είναι ο καλύτερο μηχανισμό για να το επιτύχουμε. Ο κύριο Σταυρακάκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να επικροτήσω την άμεση ενέργειά σας και να, να συμφωνήσω με τα σημεία που τονίσατε στην πρώτη σας ε, τοποθέτηση καθώς και με τα περισσότερα σημεία που έχουν τεθεί και έχουν αναφερθεί από τους ε, συναδέλφους. Ε, για μας προσωπικά θα ήθελα και θα σας παρακαλούσα αν μπορείτε στα σημεία της ε, προφορικής ερώτησης να συμπεριλάβετε δύο κέρια κατά τη γνώμη μου σημεία. Πρώτον, η πολιτική συνοχή δεν μπορεί να γίνεται με διακριτό τρόπο στην Ευρώπη. Τι θέλω να πω. Δεν πρέπει να, πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις περιφέρειες και όχι για κάποιες χώρες. Και δεύτερον, όλοι μας γνωρίζουμε ότι οι πολιτικοί συνοχή για να είναι αποτελεσματικοί θα πρέπει να εμπλέκονται ουσιαστικά και οι τοπικοί παράγοντες της περιφερειάρχης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Κρέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση. Θα συμφωνήσω με τις επιθυμίες των συναδέλφων. Θεωρώ πραγματικά απίστευτη την μέθοδο που διάλεξε ο Πρόεδρος της Επιτροπής και από άποψη ουσίας και από άποψη διαδικασίας. Διότι η Επίτροπος η οποία εργάστηκε ωστόσο επί μια πενταετία ε, στην Κομισιόν για τα θέματα αυτά απεχώρησε από την Κομισιόν έγινε Ευρωβουλευτής και ο ασκών καθήκοντα επίτροπο τώρα, ο οποίο δεν θα έχει και παραπάνω μάλλον θητεία εκεί, δηλαδή θα ασκήσει μόνο τα καθήκοντά του για αυτό το μικρό διάστημα, είναι άγνωστο ποιος θα αναλάβει στο μέλλον το χαρτοφυλάκιο αυτό και έρχεται τώρα η Επιτροπή αυτή με αυτόν τον Επίτροπο και με αυτόν τον Πρόεδρο να υποβάλει αυτή την πρόταση η οποία πρόταση ανατρέπει απολύτω τα όσα θεωρεί ή τουλάχιστον η δική μου πολιτική ομάδα ότι πρέπει να αποτελούν την πολιτική συνοχής. Δεν θεωρώ, μάλλον έχω αμφιβολίες για το αν μια προφορική ερώτηση μπορεί να είναι επαρκής. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι μόνο το πρώτο βήμα και πρέπει σύντομα να διασαφίσουμε προς ποια κατεύθυνση επιθυμεί να κινηθεί το ίδιο το Κοινοβούλιο. Για μένα είναι σαφές ότι ποτέ δεν θα μπορέσουμε να εξαιρέσουμε τα θέματα της προστασίας του κλίματος από την πολιτική της συνοχής. Κάπου εντάσσεται στην πολιτική συνοχής. Αλλά η πολιτική συνοχής για το μέλλον δεν μπορεί να εφαρμόζεται μόνο σε ένα τμήμα ε, των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής και τα υπόλοιπα να γίνονται τομιακά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ε, δίνοντας κάποια δισεκατομμύρια για την προστασία του κλίματος έχουμε εξαντλήσει και τα θέματα της πολιτικής συνοχής. Η δική μας τουλάχιστον πολιτική ομάδα έχει απολύτως διαφορετικές θέσεις από αυτές που διαλαμβάνει το έγγραφο. Άλλωστε το Κοινοβούλιο είναι ο συνομοθέτης και μετά από την σημερινή απόφαση που έλαβε το Τσεχικό Συνταγματικό Δικαστήριο θεωρώ ότι θα τεθεί σε ισχύ σύντομα η συνθήκη της Λισαβόνας και επομένως θα είναι το ε, Κοινοβούλιο συνομοθέτης σχεδόν σε όλους τους τομείς. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι τα πράγματα δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν έτσι, ότι πρέπει να υποστηριχτεί η νομοθετική εργασία και όταν πρόκειται για τη δημοσιονομική προοπτική, όπου να συμμετάσχει η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και με τα, προσώπα, με που θα ορίσει και όχι απλώς να μας θέτουν υπόψη ένα έγγραφο το οποίο μετά εμείς πρέπει να δεχθούμε. Ο κύριος Κυριλόφ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω γιατί τα είπαν οι προηγούμενοι. φαίνεται ότι ομόφωνα σχεδόν αντιδρούμε με το, στο, προς το έγγραφο αυτό της Κομισιόν. Θα ήθελα απλώς να προσθέσω το εξής. Είναι πολύ περίεργο, αλλά έχω το αίσθημα ότι γενικά κυκλοφορεί εδώ και αρκετό καιρό ότι κάποιος θέλει να αλλάξει την πολιτική συνοχής. ακούγεται, ακουγόταν και πρέπει να δούμε το θετικό σε όλα αυτά. Επιτέλους όλα αυτά συγκεκριμενοποιούνται οι φήμες. Αυτό είναι θετικό. Και είναι επίσης θετικό ότι η Επιτροπή μας τόσο ομόφωνα δέχεται να αντιδράσει. Διότι περίεργο είναι Όλοι λένε, τουλάχιστον δημόσια, ότι η πολιτική συνοχή είναι επιτυχής. Ότι καθόλου αυτά τα χρόνια που εφαρμοζόταν ήταν επιτυχής. Βέβαια όλα αλλάζουν, δεν λέω πάντα ρί. Αλλά οι κεντρικές ιδέες πρέπει να παραμείνουν άμα είναι επιτυχής. Αλλιώς δεν καταλαβαίνω διότι η συνοχή σημαίνει αλληλεγγύη και αλληλεγγύη στην Ένωση είναι κάτι που χρειάζεται επιγόντως γιατί μόνο έτσι υπάρχει μια συνεπής Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως θα έπρεπε στο τέλος κυρία Πρόεδρε να μας πείτε εσείς δεν είχατε αυτή την εντύπωση ότι κάποιος ή κάποιοι εδώ και καιρό προσπαθούν να αλλάξουν τα πράγματα. Τέλος πάντων επαναλαμβάνω ότι και εγώ υποστηρίζω όλα όσα είπαν οι προηγούμενες πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ αλλά τελειώνει ο χρόνος μας γιατί έχω ακόμη μακρύ κατάλογο κλείνει τώρα. Αν θέλει κανείς να το πει τώρα. Αν ε, έχουν υποθεί αυτά που θέλετε να πείτε παραλείπτε τα παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος αν και το θέμα ε, είναι ευρύ. Το θέμα των σχέσεων δηλαδή μεταξύ Κομισιών και Ευρωπαίου πολίτη. Ακούσαμε ορισμένα πράγματα ήδη από την πράσινη λεγόμενη βίβλο που ήταν ασαφής και καθόλου συγκεκριμένη ως προς το μέλλον για τη συνοχή. Όπως είπε και ο συνάδελφος Ευγένιος προηγουμένως, Κύριλοφ, όντως κάτι ακουγόταν, φήμες ακούγονταν και ο πρόεδρος της Κομισιόν όταν συνάντησε όλες τις πολιτικές ομάδες δεν έκανε την παραμικρή νήξη για τις προθέσεις του αλλαγής της περιφερειακής πολιτικής. Ούτε γενικά καν δεν την ανέφερε, την πολιτική συνοχή μάλλον. Και πιο συγκεκριμένα η Κομισιόν που βρίσκεται στο τέλος της θητείας της ξαφνικά έρχεται να μας υποβάλει μία ριζική αλλαγή αλλά με ποια πολιτική και δεοντολογική βάση υπήρξε διαπραγμάτευση μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου όχι υπήρξε διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο ούτε φαντάζομαι με τι ενθουσιασμό οι χώρες σε εισαγωγικά οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης τα ακούν όλα αυτά. Πώς ε, τολμάει η Κομισιόν να προτείνει ένα τέτοιο έγγραφο ενώ αναμένεται ακόμα η έγκριση από το, από το Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο εάν με τέτοιες μεθόδους ελπίζουν να εφαρμόσουν τη μελλοντική πολιτική συνοχή, τότε δεν πρέπει να περιμένουν τίποτα. Και ελπίζω να συμφωνήσουμε όλοι από αυτού. Αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο βρίσκεται ενώπιον τετελεσμένου γεγονότος ή επιχειρείται ένα τετελεσμένο γεγονός. Θα ήθελα να πιστεύω ότι εμείς εδώ στην Επιτροπή μας είμαστε σε θέση να γράψουμε ένα έγγραφο που να ορίζει τις ιδέες μας και τις προθέσεις μας με την υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Γιατί ε, αυτό θα ήταν μια πραγματικά σοβαρή πολιτική κίνηση που να τη λάβει υπόψη της η μελλοντική Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μην μπορέσει δηλαδή να αλλάξει τις βάσεις της περιφερειακής πολιτικής προς κατευθύνσεις που θα θέσουν εν κινδύνο την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Κύριε κύριος Λάστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διάβασα το σχέδιο της ανακοίνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το παρουσιάζει ως βάση μια συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις ε, μελλοντικέ δημοσιονομικές προοπτικές και με ανησυχεί το γεγονός ότι περιλαμβάνονται σκέψεις ε, για την πολιτική συνοχή, οι οποίες πόρο απέχουν από τις θέσεις της Επιτροπής μας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει λοιπόν να επενθυμίσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον βασικό ρόλο των περιφερειών για τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο έγγραφο όπως είναι η ανάπτυξη και η απασχόληση, όπως επίσης και η προστασία της ε, ε, του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Με ενδιαφέρουν επίση και οι μεταβατικέ περίοδοι που αναφέρονται στο κείμενο και το γεγονό ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το στόχο τη ανταγωνιστικότητα. Επίση, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι με την επικύρωση τη συνθήκη τη Λισαβόνα, ε, η πολιτική συνοχή θα είναι μια εγκάρσια πολιτική ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, από κοινού με την κοινωνική και οικονομική πολιτική. Ο κύριος Φρανς Όμπερμαϊτ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ταχύτατη αντίδρασή σας ε, στην, στο έγγραφο. Είμαι νέο μέλος στην Επιτροπή και πραγματικά μένω κατάπληκτος, διότι όποιος συνέταξε την πρόταση αυτή, προφανώς κάτι σκεφτότανε. Δεν, δεν μπορώ να υποθέσω ότι πρόκειται για κανένα καλαμπούρι, αλλά έχοντας ήδη στις πρώτες εδώ συνεδριάσεις ακούσει πολλά θετικά υπέρ της περιφερειακής πολιτικής, βλέπω εδώ να γίνεται στροφή 180 μοιρών. Και για πραγματικά, πρόκειται πραγματικά για μια καρικατούρα πολιτικής. Κατ' εμέ πρέπει να απορριφθεί η πρόταση. Από κάθε άποψη. Είναι επίσης απογοητευτικό για όλους όσοι άκουσαν τις ωραίες πανηγυρικές ομιλίες ε, στις ε, ε, πρώτες συνεδριάσεις με τους προέδρους κτλ. Θα είναι πολύ απογοητευμένοι ακούγονται. Φεύγουμε από εδώ, επιστρέφουμε στις χώρες μας και θέλουμε να μπορέσουμε να διηγηθούμε στους ψηφοφόρους μας θετικά πράγματα με την σχεδιαζόμενη στρατηγική για το χώρο του Δούναβη και ούτω καθεξής. Και τώρα γίνεται προσπάθεια να κατατμηθεί σε, σε τομείς. Με την πολιτική αυτή, με την πολιτική αυτή, με την εδώ την πρόταση, δεν προσφέρουμε απολύτως καμία θετική υπηρεσία στην Ένωση. Και σίγουρα δεν πρόκειται να αλλάξει η διάθεση του ευρωπαϊκού κοινού απέναντι στην ε, κοινότητα και στην Ένωση με τέτοια πράγματα. Η κυρία Μπόμπινσκα. Νομίζω ότι στη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πραγματικές διαφορές στην Ευρώπη και ποια είναι η εικόνα που δίνει σήμερα η Ευρώπη. Όχι μόνο υπάρχουν τα 10 νέα μέλη, αλλά ακόμα πιο ε, πρόσφατα ε, με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και θα μπουν και άλλες νέες χώρες μέλη που επίσης δεν είναι πλούσιες. Οι δε περιφερειακές διαφορές στην Ευρώπη θα γίνουν ακόμα πιο έντονες από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο θέλουμε να επανορίσουμε την περιφερειακή πολιτική. Δεύτερο, πρέπει να εξετάσουμε την ε, πολιτική της Λισαβόνας. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για περιφερειακή πολιτική αν δεν συζητήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ως στόχο, ε, να, μάλλον τους ίδιους παρόμοιους στόχους. Είναι λοιπόν αποτελεσματική η στατική της Λισαβόνας ή όχι. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι δεν είναι αρκετά αποτελεσματική. Πρέπει να αναθεωρηθεί λοιπόν, να εξεταστεί, να επανεξεταστεί εδώ στην Επιτροπή μας. Πρέπει να εξετάσουμε όλα αυτά τα μέτρα και τους μηχανισμούς που ακολουθούν τους ίδιους σκοπούς και εάν αποδειχθεί ότι κάποιο, κάποιος μηχανισμός δεν είναι αποτελεσματικός πρέπει να δούμε, εάν τον αφήσουμε, να τον εγκαταλείψουμε, ποιος θα είναι αποτελεσματικός. Ένα τρίτο επιχείρημα κατά μιας νέας κατεύθυνση είναι το εξή. Βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσεως. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς αυτή, τι επιπτώσεις θα έχει αυτή στις περιφερειακές διαφορές. Χρειάζεται λοιπόν να λάβουμε υπόψη τον παράγοντα αυτό στην διατύπωση, συζήτηση και διατύπωση της νέας περιφερειακής πολιτικής. Εάν η κρίση οδηγήσει σε βάθεμα των διαφορών, δεν μπορούμε να αφήσουμε να χαθεί ένας μηχανισμός ο οποίος στηρίζει την ε, περιφερειακή συνοχή. Σοφή Μπριά. κυρία Πρόεδρε. Εκφράζω και εγώ την ικανοποίησή μου για την ε, απάντηση που δώσατε στην πρόταση, για την αντίδρασή σας δηλαδή. Και όντας και εγώ νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, δηλώνω και εγώ την ε, από πλευράς μου απόρριψη του εγγράφου αυτού που υπάρχει και δεν υπάρχει και για την ουσία και για την μέθοδο. Η κρίση σήμερα πλήττει όλες τις χώρε μέλη της Ένωσης και περισσότερο από ποτέ κάθε χώρα μέλος έχει ανάγκη από μια πολιτική συνοχής. Το σημείωμα αυτό που υπάρχει ή δεν υπάρχει και που μας απευθύνεται σήμερα μέσα σε περίοδο οικονομικής και κοινωνικής κρίσης είναι απολύτως απίστευτο. Η πολιτική των περιφερειών δίνει ένα πραγματικό πρόσωπο στην Ευρώπη. Είναι ένας μηχανισμός που μας επιτρέπει να δώσουμε συγκεκριμένη μορφή σε δράσεις και δεν πρέπει να έχει χαρακτήρα αποκλεισμού. Οι χώρες που αναπτύσσονται οικονομικά έχουν ανάγκη από αυτή την πολιτική κοινωνική συνοχής και οι άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η χώρα μου δηλαδή, βρίσκονται μέσα σε μια, οικονομική, σε μια φάση οικονομικής μεταμόρφωσης κατά τη θεωρία του Σλουμπέτερ που έχει ένα δημιουργικό χαρακτήρα και χρειάζεται όμως υποστήριξη ώστε τα κράτη να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια που κάνουν και οι επιχειρήσεις σε μια μεταρρύθμιση, μια μεταμόρφωση. Όπως είπε και ο συναδελφός μου Γιάνν Ολμπριχτ, πρέπει από τώρα να αρχίσουμε να εργαζόμαστε επί προτάσεων που θα είναι τέτοιες που να απαντήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Σαγκουράκης παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ως ε, νέο μέλος και εγώ της Επιτροπής θα ήθελα να εκφράσω την αγανάκτηση και την ε, σοβαρή καταγγελία για αυτό το έγγραφο που κυκλοφορεί. Πολύ φοβάμαι ότι επίτηδες υπάρχει αυτή η διαρροή. Πολύ φοβάμαι ότι η Επιτροπή έχοντας υπόψη ότι ασφαλώς ότι η κρίση θα εντείνει και θα οξύνει ακόμα περισσότερο τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών, μας προετοιμάζει από τώρα για το τι πρόκειται να γίνει. Επίσης, κυρία Πρόεδρε, εμένα δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση τη στιγμή που έρχεται αυτό το κείμενο. Έρχεται τη στιγμή που ε, μετά από εκβιασμούς και πιέσεις ο λαός της Ιρλανδίας τελικά ε, επικύρωσε τη συνθήκη της Λισαβόνας έρχεται αμέσως μετά την επικύρωση και από την Τσεχία και είναι σαν να μας λέει η Κομισιόν, ξέρετε κάτι, τώρα σας έχω στο τσεπάκι μου και σας κάνω ό,τι θέλω. Κλείνοντας, πολύ φοβάμαι ότι αυτό το πράγμα έχει βγει στη δημοσιότητα ώστε προφανώς και να αντιδράσουμε και να αντιδράσουμε με δρυμύτατο τρόπο μετά να μας φέρουν μια δεύτερη εκδοχή η οποία θα είναι λίγο καλύτερη να μας πούν ότι πήραν υπόψη τους ε, την κριτική μας και έτσι τελικά να περάσει αυτό το σχέδιο που θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερες ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω σχεδόν καλυφθεί σε αυτά που θέλω να πω. Τρία σημεία θέλω να τονίσω. Πρώτον, δεν είναι χωρίς βάση και αιτία η ανησυχία εκφράστηκε σήμερα. Κατά διαστήματα έρχεται μια τέτοια άποψη για μια νέα περιφερειακή πολιτική. Δεύτερον, ότι είναι σαφές από, τις, από αυτά που υπόθηκαν σήμερα ότι το Κοινοβούλιο επιμένει σε μια περιφερειακή πολιτική που είναι συμφασμένη με τη φύση της Ένωσης και με τις αξίες αλληλεγγύης. Και τρίτον, θα ήθελα να τονίσω και εγώ ότι πρέπει αυτό να συνδεθεί με την οικονομική κρίση και με την ε, με την ανησυχία για το ότι η ανάκαμψη δεν φέρνει θέσεις απασχόλησης. Λοιπόν, νομίζω ότι εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Δεν είμαστε Επιτροπή Απασχόλησης, αλλά οι θέσεις εργασίας είναι άμεσα συνειφασμένες με το δυναμισμό που μπορούν να αναπτύξουν οι περιφέρειες και πρέπει αυτό να μας απασχολήσει ιδιαίτερα και στο πλαίσιο αυτό και στο πλαίσιο, όπως είπε η συνάδελφος, της αναθεώρησης στρατηγικής της Λισαβόνας. Σας ευχαριστώ πολύ. The last very short statement, Mr. Goodmanis, please. Very short. Um, when we when when when we step in the shoes of Commission. Εάν προσπαθήσουμε να παίξουμε τον ρόλο της Κομισιόν, θα δούμε ότι δεν είναι και ορκισμένοι εχθροί της περιφερειακής πολιτικής. Το έγγραφο ίσως εμφανίστηκε με τον τρόπο αυτό για δύο λόγους. Αφενός μπορεί να τους ανησυχεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο, στην παγκόσμια σκηνή και να λένε ότι οι πολιτικές δεν αποδίδουν. Και στην περίπτωση όπου το ε- ευρώ πρέπει να ανταγωνίζεται. Καλά, ανταγωνίζεται και με άλλες περιφέρειες ή κράτη. Το ερώτημα είναι εάν δαπανούμε πολλά χρήματα για να αναπτύξουμε ισοδύναμα τις διάφορες περιφέρειες εγώ είμαι σαφώς μέλος από τι ε, νέες χώρες και ε, ψηφίζω και με τα δύο χέρια υπέρ της πολιτικής συνοχής, αλλά αυτή ε, η εξίσωση ίσως να μην συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και ίσως αυτός είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο μιλούν για τομεακή αντιμετώπιση και το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι σε περιπτώσεις κρίσεων οι χώρες, οι χώρες ενδεχόμενα να προσπαθήσουν περισσότερο να ανακτήσουν κάποιες ευθύνες. Δεν αρκεί βέβαια να ασκείται κριτική. Πρέπει και εμείς να ε, συμβάλλουμε με κάποιες αντιπροτάσεις ενδεχομένως. Δείχνοντας και η δική μας στάση για να βελτιώσουμε την ε, ε, περιφερειακή ανάπτυξη και την εξίσωση του επίπεδου, του βιωτικού επίπεδου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, η Επιτροπή να θέλει να μας προκαλέσει λίγο να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Πρόεδρος. Όλα αυτά ήταν η ε, βασική αντικειμενική στόχη της προηγούμενης περίοδου και ε, να περάσει και η Λισαβόνα στο περιφερειακό επίπεδο, μέχρι εκεί δηλαδή. Αλλά και πολλά έχουν γίνει. Δεν μιλούμε όμως τώρα για την πολιτική της δεκαετίας του 80, αλλά για τις πολιτικές του 2006, που είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είχαμε ε, πριν από 20 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάντως όλες και όλους για τα σχόλιά σας, που ήταν πάρα πολύ χρήσιμα. Όλες οι παρεμβάσεις σας ήταν πολύ χρήσιμες ε, Μαθαίνω ότι υπάρχει μια συμφωνία για την υποβολή προφορικής ερώτησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ίσως θα χρειαστεί να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε μεταξύ των συντονιστών για το ποιες ερωτήσεις, ποιες θα είναι οι βασικές ερωτήσεις που θα περιλάβουμε. Γιατί θα πρέπει να είναι προφορική ερώτηση επί της ουσίας και όχι επί πολιτικών και διαδικασιών. διαδικασιών. Αυτό ε, καταλαβαίνω ότι είναι και η δική σας θέση και συμφωνεί με τη δική μου. Ορισμένοι από εσάς Είπατε επίσης ότι πρέπει η Επιτροπή Ρέτζι το δυνατόν συντομότερο να καταθέσει τη δική της συνολική θέση. Οι συντονιστές θα εξετάσουν σήμερα την πρότασή μου να φτιάξουν μια ομάδα εργασίας μέσα στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης με εκπροσώπους όλων των πολιτικών ομάδων για να εξετάσουν τη μελλοντική πολιτική συνοχής και ελπίζω ότι μπορούμε να κάνουμε συζήτηση αυτή και για την προφορική ερώτηση και να ε, φτιάξουμε και αυτή την ομάδα εργασία, η οποία ε, θα συζητήσει τα θέματα αυτά το δυνατόν συντομότερο. Αν με επιτρέπετε λοιπόν θα ε, θεωρήσω ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το θέμα αυτό. Ελπίζω ότι οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ήδη παρόντες και μπορούν να μας Okay, so we move now to, okay. So we move now... Καλά, προχωρούμε... στην ε, πρόταση της κυρίας Κάρη Μαντελή για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Θα ενθυμίσετε ότι είχαμε ήδη κάνει μια ανταλλαγή απόψεων για τη γνωμοδότηση. Στο μεταξύ αρμόδια επί επιτροπή, ναι, I just stop for 20 seconds to... Θα περιμένω για λίγο για να μπορέσετε να αποχωρήσετε. Take the seats. Still I would like to ask you to do it as fast as possible. Παρακαλώ μου σύντομα. Να σας πω ότι η ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Πολιτισμού άλλαξε που είναι αρμόδια για ε, το έτος εθελοντισμού και πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα της ατζέντα και γι' αυτό βάλαμε σήμερα στην ημερήσια διάταξή μας το θέμα αυτό για ε, την πρόταση αποφάσεως του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού και θα παρακαλέσω την κυρία Καρή Μαντέλη να αναπτύξει τις θέσεις της για τις τροπολογίες. Γιατί είχαμε και προθεσμία, έχουν κατατεθεί 20 τροπολογίες. Άρα, ε, σύντομα κυρία Ντέλη και παρακαλώ να μου ε, πείτε και τα σχόλιά σας επί των τροπολογιών. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προηγούμενους συναδέλφους για τη δουλειά τους που μας επέτρεψαν το 2011 να γίνει το έτος εθελοντισμού. Επίσης σας ευχαριστώ υπάρχοντα τωρινά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τις προτάσεις τροπολογιών που καταθέσατε και που βελτιώνουν τους στόχους του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι θεωρώ ότι όλες οι τροπολογίες εμπλουτίζουν το κείμενο και προσθέτουν απαραίτητα στοιχεία σε αυτό για να γίνει το έτος εθελοντισμού επιτυχές. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ στο γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο, κλίμα μέσα στο οποίο εξετάζουμε το θέμα μας. Στην προηγούμενη συνεδρίαση θα θυμάστε της Επιτροπής Περίφ είχαμε μόλις μάθει τον ορισμό του εισηγητή κυρίου Μάρκος Κούρια της Επιτροπής Πολιτισμού. Για να υπάρχει περισσότερη και ακριβέστερη δεοντολογία και διαφάνεια πρέπει να σας πω ότι πριν από 10 μέρες έγινε στο Στρασβούργο μία συνάντηση με το σύνολο των εισηγητών και σκιωδών όλων των επιτροπών και όλων των πολιτικών ομάδων. Και τότε είδα στη συνεδρίαση εκείνη ότι υπήρχε, προβλεπόταν μία επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος για να προλάβει η Σουηδική Προεδρία. Γι' αυτό τόνιζα πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος και η εργασία των χνομοδοτικών επιτροπών που είναι πάντοτε σοβαρός και ανταποκρίνεται στην εικόνα και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως νέο μέλος του θα ήθελα κύριοι συνάδελφοι να τονίσω ότι η διαδικασία που επελέγει ήταν ε, δεν αντίθετη με τη θέλησή μου. Αντί να περιμένουμε, χρειάστηκε δηλαδή να σημειωθεί μια καθυστέρηση για να περιμένουμε το αποτέλεσμα της έγκρισης της Λισαβόνας και μετά ξαφνικά άλλαξε η στάση και ζητήθηκε επιτάχυνση μετά τις καθυστερήσεις ιδιαίτερα από την Επιτροπή Απασχόλησης και Προϋπολογισμού. Όλα αυτά για να ικανοποιηθεί η βιασύνη της, ε, η έλλειψη χρόνου της Σουηδικής Προεδρίας. Στο Στρασβούργο επίσης μας πρότειναν νέα διαδικασία για τις τροπολογίες χωρίς εσείς κύριοι συνάδελφοι και των υπολείπων επιτροπών να έχουν μπορέσει να τις μάθουν. Εγώ ανέμενα ως νέα Ευρωβουλευτής με γιώτα επειδή δίνω σημασία στη δουλειά μας και στις απόψεις σας που βελτιώνουν τα κείμενα περίμενα και περιμένω σήμερα να αναλύσουμε μαζί από κοινού τις τροπολογίες. Για μένα είναι ουσιώδες η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης να μπορέσει να γνωμοδοτήσει όπως πρέπει ώστε με φιλόδοξους στόχους το έτος εθελοντισμού 2011 να γίνει ένα εργαλείο για την προώθηση του ε, χαρακτήρα της ευρωπαϊκής Ιθαγένειας και της αλληλεγγύης. Γι' αυτό αγαπητοί συνάδελφοι μελέτησα καλά τις τροπολογίες σας και νομίζω όπως το είπα και πριν ότι εμπλουτίζουν το αρχικό κείμενο γιατί αυξάνουν κονδύλια, αυξάνουν την προστασία των εθελοντών ή προσθέτουν αξία στη δουλειά τους. Είμαι λοιπόν πολύ ικανοποιημένη από τις τροπολογίες και δεν έχω να προσθέσω τίποτα ουσιαστικό. Μόνο μία αποσαφηνισούλα για μια τροπολογία του κυρίου Κίλη όπου θα ήθελα η λέξη delinquency να αντικατασταθεί από τη λέξη idleness σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας, για αυτή τη δουλειά που κάνατε και ελπίζω ολόψυχα οι συζητήσεις μας να έχουν αποτέλεσμα και για την Επιτροπή Παλιτισμού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντελή. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει το λόγο. Yes, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την κυρία Ντελή, γιατί εργάστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Χρειάστηκε όλοι να επιταχύνουμε λίγο για να προχωρήσει το θέμα. Και να πω ότι καλωσορίζω και τις τροπολογίες της, οι οποίες ε, έχουν ε, δημιουργήσει μια πιο στεναρή εικόνα για το έγγραφο. Και εγώ είμαι νέα Ευρωβουλευτή και νομίζω οι περισσότεροι από εμά που καταθέσαμε τι τροπολογίε είμαστε νέοι. Και όχι μόνο χρειάστηκε να εργαστούμε γρήγορα, χρειάστηκε να εργαστούμε και πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύαμε. Ναι. Έχω κάνει και εγώ κάποιες τροπολογίες και με χαρά διαπιστώνω ότι οι τροπολογίες της κυρίας Δελή ε, παρουσιάζουν μια πιο επαγγελματική προσέγγιση για τον εθελοντισμό και θεωρούμε ότι το έτος εθελοντισμού είναι η χρονιά η οποία θα μας επιτρέψει να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικέ ε, πρακτικές μεταξύ κρατών μελών. Υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ναι. μακρά παράδοση εθελοντισμού και έχουν πρακτικές και κάποιες άλλες οι οποίες μόλις μπαίνουν στη διαδικασία και αντιμετωπίζουν ίσως το θελοντισμό με άλλο τρόπο. Αυτό που προσπάθησα να κάνω εγώ με τις ε, τροπολογίες μου είναι να εισαγάγω ένα σύστημα πιστοποίησης. διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται ως θελοντές και θα ήθελαν να περάσουν σε επαμοιβή εργασία και ίσως κάπου θα πρέπει να αναγνωρίζεται και η δουλειά τους ε, και να μην θεωρούνται ότι ε, δεν κάνουν κάποια δουλειά που δεν έχει αξία επειδή είναι εθελοντές. Ε, να μπορεί δηλαδή ο μελλοντικός του εργοδότης να αναγνωρίζει ότι υπάρχουν κατάλληλες πρακτικές, να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση, κατάρτιση και να υπάρχουν διάφορες πρακτικές που ξέρουν ότι πρέπει να δίνουν οι εργοδότες και ελπίζω ότι μέσω συζητήσεων και μέσω συναντήσεων με άλλους οργανισμούς ε, κατά το έτος εθελοντισμού θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε τα θέματα αυτά. Ε, η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ που παρουσιάσετε το θέμα των βέλτιστων πρακτικών, διότι είναι ένα από αυτά τα οποία δεν έχουμε εκμεταλλευτεί ακόμα επαρκώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κέλλη. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ είμαι νέος Ευρωβουλευτής και χαίρομαι που συμμετέχω ω και όδηση σε αυτή τη γνωμοδότηση. Νομίζω ότι ο εθελοντισμός είναι ένας από τους μεγάλους στόχους του ανθρωπίνου είδους, από αυτούς που μας διαχωρίζει από το ζωικό βασίλειο, το γεγονός ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε κοινότητες και ε, χαίρομαι για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει ένα ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού. Από την ημέρα που εμφανίστηκα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακούω παντού την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο κοντά στους πολίτες της. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού είναι μια τέτοια ευκαιρία. Παρουσίασα και εγώ κάποιε τροπολογίε, μικρέ αλλαγέ, δεν ε, είναι ρηξικέλευτε οι αλλαγέ, διότι η γνωμοδότηση τη κυρία ε, Ντέλη και οι τροπολογίε τη είναι εξαιρετικέ. Έχω εστιάσει κυρίω στον τομέα του αθλητισμού διότι με την ε, θέση εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας ε, είναι πολύ σημαντικό να αντικατοπτρίζεται αυτό και σε όλους τους τομείς και από τη χώρα μου, από την Ιρλανδία, γνωρίζω από μία έκθεση ότι το 50% των ανθρώπων που εργάζονται εθελοντικά είναι στον τομέα του αθλητισμού. Επομένως θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους εθελοντές ε, στον τομέα αυτό. Ε, φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και κάποιες συμβιβαστικέ τροπολογίε, αλλά νομίζω ότι μπορούν να λυθούν τα προβλήματα και δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τη γνωμοδότηση. Ε, να πω γιατί είμαστε κατά κάποιων τροπολογιών. Καταρχήν για την τροπολογία 7. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι απαραίτητη η ε, τροπολογία αυτή, διότι ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδεύουμε προς την κατεύθυνση της ε, παροχής υγείας για όλους. Ο Πρωθυπουργό ε, Μπέρτι Άχερν στην ε, χώρα μου δημιούργησε μία ομάδα για να συζητήσει για τα θέματα αυτά και ε, οι περισσότεροι από τους εθελοντές ασχολούνται με το θέμα του κόστους της ασφάλισης υγείας. Και αυτό είναι ο αναποτρεπτικός παράγοντας. Επίσης πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εθελοντέ θα μπορούν να εργαστούν με πλήρη απασχόληση και τα έξοδά του θα πρέπει να αποζημιώνονται. Ναι, μεν συμφωνούμε με αυτό, αλλά άτομα τα οποία εργάζονται με πλήρη απασχόληση και προσφέρουν και θελοντικό έργο, Ορισμένε φορέ μπορεί να πρέπει ένα επαγγελματία να αντικαταστήσει με ένα εθελοντή. Δεν γίνεται πάντα αυτό και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση. Πολλοί από του εθελοντέ πολλέ φορέ δεν ζητούν καμία αποζημίωση για τα έξοδα του. Ε, υπάρχει ένα από του πολύ μεγάλου αθλητέ στην Ιρλανδία που 50 χρόνια προσέφερε έργο και δεν ζήτησε ποτέ αποζημίωση. Δεκάρα τσακιστή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Καταλαβαίνω πώς προκύπτει η τροπολογία. Ε, λέμε ότι πρέπει να δαπανούνται χρήματα για διαφημιστικές εκστρατείες, αλλά νομίζω ότι δεν μας το επιτρέπει το κόστος και νομίζω ότι ε, δεν θα επιτύχουμε και πάρα πολλά. Για να επανέλθω και πάλι στη δική μου πείρα με αυτή την ομάδα που σας ε, ανέφερα και πριν, οι περισσότεροι από τους εθελοντές δεν το κάνουν γιατί τους το ζητάνε. Ο λόγος για τους οποίους είμαι εγώ σκιώδης εισηγητές, για παράδειγμα εδώ, ε, είμαι σκιώδης γιατί μου το ζήτησε ο κύριος Βανίστερ Λορόι και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ κύριο Σόβερμαϊ. Pardon? Microphone? Does it work Okay. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αξίζει έπαινος ε, στην ε, εκπόνηση του έργου αυτού. Προέρχομαι από μια χώρα, την Αυστρία, η οποία έχει την υψηλότερη πυκνότητα εθελοντών. 60% των Αυστριακών ασχολούνται με τέτοια θέματα. Είναι σημαντικά αυτά που γράφει ε, το έγγραφο. Συμφωνώ και με τον προαναλύσαντα. Βέβαια, από την άλλη μεριά η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι σαφή. Όπως για παράδειγμα για τους πυροσβέστες ή για τους διασώστες υπάρχουν και φαιές ζώνες όπου η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι δεδομένη. Διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι και επαγγελματίε και ε, εγκαταλείπουν τα επαγγέλματά τους για να ασκήσουν ε, τις εθελοντικές υπηρεσίες. Πρέπει εδώ να ε, γίνει μια πρόταση να υπάρξουν ενιαίες ρυθμίσεις. Επίσης, τα σχετικά με την περίθαλψη είναι σημαντικό για τέτοιες οργανώσεις που, επαναλαμβάνω, όπως στην περίπτωση των πυροσβεστών ή των διασωστών, ε, θέτουν σε κίνδυνο και την υγεία και την ζωή τους καμιά φορά, Χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρξει ρύθμιση για ε, θέματα υγείας και κυρίως για να περνούν από εξετάσεις κλπ. Μάρκος Κούρια, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι αναπληρωτής εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά επειδή είμαι και ο εισηγητής στην Επιτροπή Πολιτισμού για το θέμα αυτό, θεωρώ ότι θα πρέπει να παρέμβω. Καταρχήν για να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Καρή Μαντελή για το έργο της και μαζί με αυτήν και όλους ε, εσάς εδώ στην Επιτροπή διότι οι τροπολογίες που παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Όπως σας υπενθύμησε και η ίδια συνάδελφος, ε, συναντηθήκαμε στο Στρασβούργο και με όλα τα μέλη των ενδιαφερομένων επιτροπών προκειμένου να μπορέσουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού να είναι κάτι το οποίο θα είναι όσο το δυνατόν ε, κοινό και να μπορέσουν να συμμετέχουν ενεργά όλες οι επιτροπές που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Η συνάδελφος πριν σας ε, υπενθύμησε πόσο γρήγορα πρέπει να εργαστούμε για αυτό το θέμα και εδώ θα ήθελα ε, να εξηγήσω λίγο καλύτερα τι ακριβώς γίνεται, διότι αλλιώς ε, ελοχεύει ο κίνδυνος να είναι περίπλοκα τα πράγματα και να μην κατανοήσουμε γιατί τόση βιασύνη. Δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο που αφορούσε στη Σουηδική Προεδρία. Το βασικό πρόβλημα είναι η νομική βάση επί της οποίας ε, αποφασίζεται αυτό το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού και κυρίως το όλο θέμα που αφορά στην πιθανή ε, θέση σε ισχύ της συνθήκης ε, της Λισαβόνας. Βάσει των νομικών μας υπηρεσιών, με την θέση σε ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνας, εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούμε απλά να γνωμοδοτήσουμε για αυτό που θα μας παρουσιάσουν. Θα μπορούμε απλά να πούμε λοιπόν αν το κείμενο που μας παρουσιάζεται μας αρέσει ή όχι. Ο περιορισμός μας λοιπόν είναι να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε ένα κείμενο. Επειδή λοιπόν όλοι θέλουμε να μεριμνήσουμε ώστε ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια τέτοια διαδικασία ε, να είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Συνεργαστήκαμε λοιπόν, μιλήσαμε και με εκπροσώπους του Συμβουλίου αλλά και με τον αρμόδιο επίτροπο για να δούμε Εάν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εργασία αυτή πριν από το τέλος του έτου, το έτους υπάρχει και μια ε, σχετική βιασύνη γιατί μπορεί να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας από 1η Ιανουαρίου. Αποφασίσαμε λοιπόν, δεδομένου ότι έχουμε εργαστεί από κοινού για το θέμα αυτό, να βιαστούμε λίγο για να δοθεί και αξία στα όσα έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, μεν λοιπόν υπάρχει αυτή η βιασύνη, αλλά υπάρχει και αναγνώριση και από πλευρά του Επιτρόπου και τη ε, Προεδρία ότι μα δίνεται η δυνατότητα να εργαστούμε για το κείμενο αυτό και μέσω των τροπολογιών που θα παρουσιάσει το Κοινοβούλιο από τι διάφορε επιτροπέ θα μπορέσει να εισακουστεί και η άποψη του Κοινοβουλίου. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι πάμε λίγο επιτροχάδιν, ε, ελπίζουμε να μπορέσουμε να έχουμε ένα κείμενο στο οποίο θα είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κίνδυνος είναι, εάν καθυστερήσει πολύ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί απλά να πει ναι ή όχι στο κείμενο που του παρουσιάζεται. Γι' αυτό άλλωστε και η ε, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού απέστειλε μία επιστολή σε όλους τους πρόεδρους των αρμοδίων επιτροπών για να τους δώσει ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο γνωρίζετε και εσείς κυρία Πρόεδρε, και να εξηγήσει λίγο τους λόγους για τους οποίους ε, προχωράμε τόσο γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν τα κάνουμε όλα βιαστικά, αλλά ε, η βιασύνη οφείλεται στην ανάγκη μας να συμμετέχει ενεργά και το Κοινοβούλιο. Ε, και ως μέλος λοιπόν της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και επειδή είμαι ο αρμόδιος ε, εισηγητής ε, στην Επιτροπή Προϋπολογισμού ή, ε, στην Επιτροπή Πολιτισμού είμαι στη διάθεσή σας για να μπορέσουμε να δούμε από κοινού και με τους εκπροσώπους της Προεδρίας και με τον Επίτροπο το θέμα για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε όλα όσα κάνουν οι διάφορες επιτροπές. Ε, την επόμενη Παρασκευή θα εξεταστεί το θέμα για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού και μετά από αυτό υποθέτω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή πορεία προκειμένου να κάνουμε και τις τροπολογίες στα κείμενα που θέλουμε να κάνουμε και να καταλήξουμε και σε μια συναπόφαση παρόλο που δεν μπορούμε να την αποκαλούμε επισήμως συναπόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, εκτιμώ τα σχόλιά σας και πριν ε, δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, να πω ότι έχουμε τρεις προσκεκλημένους από την Αυστρία, την κυρία Χάιντε Μαρία Ονοντή, τον κύριο Άντων Χάινς, μέλος του Αυστριακού Κοινοβουλίου και τον Γκέρχαρ Ράσμπουρκαν, ε, μέλος του ε, Περιφερειακού Αυστριακού Κοινοβουλίου. Καλώς ορίσατε λοιπόν και ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Να συνεχίσουμε λοιπόν ο Σελβατόρες Καρόνα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να πω ότι εκτιμώ ειλικρινά τα όσα έκανε η συνάδελφος Ντελή. Μπόρεσε να ενισχύσει πολύ περισσότερο την αξία αυτού του ευρωπαϊκού έτους εθελοντισμού, το οποίο θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να το υποτιμούμε, διότι μπορεί να αποτελέσει ένα από τα ουσιαστικά μέσα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να ενδυναμώσουμε ακόμα και το θέμα της συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε γενικές γραμμές ε, νομίζω λοιπόν ότι έγινε καλή δουλειά και με τις διάφορες τροπολογίες που παρουσιάστηκαν και φρονώ ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας δεν μπορεί παρά να είναι θετική. Τα μόνα δύο στοιχεία τα οποία ίσως είναι λίγο προβληματικά είναι το γεγονός ότι εμείς με αυτή τη γνωμοδότηση ε, θεσπίζουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού και σε κάποιες ίσως εκφράσεις ε, του εγγράφου περνάμε και σε μία ρύθμιση η οποία, αν θέλετε, δεν συνάδει απόλυτα με το στόχο που συζητάμε. Σε γενικές γραμμές βέβαια μου φαίνεται ότι το μήνυμα ε, είναι απόλυτα θετικό και εάν ενισχυθεί και από αύξηση της χρηματοδότησης που προβλέπεται ε, θα μπορέσουμε να αποστείλουμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Ε, νομίζω ότι συλλογικά έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι αυτά που είπε και ο συνάδελφος Κουρία, το γεγονός ότι θα μπορέσουμε ε, ακόμα και αυτές τις λίγες εβδομάδες που απέχουν από την ε, τελική απόφαση να συνεργαστούμε, είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αγκουράκης. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω ότι πράγματι η κυρία Καρίμα Ντελή έχει κάνει μια σοβαρή δουλειά όπως ε, και προηγούμενα. Ε, φοβάμαι ότι θα σας απογοητεύσω λιγάκι, αλλά θέλω να αξιοποιήσω την ε, παρουσία μου για να βάλω δύο-τρεις σκέψεις που πιθανώς να μπορέσουν να μας βοηθήσουν στο μέλλον. Καταρχήν νομίζω ότι όλοι μας είμαστε θελοντές. Αυτό όμως δεν έχει οδηγήσει και καλώς κατά τη γνώμη μου να έχουμε ένα ευρωπαϊκό έτος των πολιτικών κομμάτων. Και στα πολιτικά κόμματα η συνεισφορά εθελοντική είναι, φαντάζομαι και στα πολιτικά κόμματα υπάρχουν οι αξίες για τις οποίες γίνεται λόγος στην έκθεση για το έτος εθελοντισμού. Το δεύτερο που ήθελα να σημειώσω. Έτσι ε, είναι. Εγώ νομίζω έτσι είναι. Αλλιώς βέβαια θα σας πω τι νομίζω ότι κρύβεται από πίσω. Το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, ακριβώς επειδή δούμε σε μια καπιταλιστική κοινωνία, έχουμε την κρίση, την ανεργία, ναρκωτικά και πάρα πολλά προβλήματα και επειδή έρχομαι και από την Ελλάδα μπορώ να σας πω ότι είναι ακόμα περισσότερο, πραγματικά χρειάζεται αλληλεγγύη, σύμπνοια, βοήθεια, εθελοντισμός. Δεν χωράει καμία αμφιβολία. Το μόνο πρόβλημα όμως που έχω είναι ότι τα κόμματα τα αστικά κόμματα, τα κυβερνητικά κόμματα δεν είναι σε θέση να προσφέρουν αυτές τις κοινωνίες. Και ακριβώς αυτό το λόγο έρχονται να καλύψουν οι εθελοντικές οργανώσεις. Και οι λεγόμενες εθελοντικές οργανώσεις, γιατί σας ρωτάω, είναι όλες οι οργανώσεις εθελοντικές. Παραδείγματο χάρη, εγώ δεν θα ήθελα στην Ελλάδα να φτάσουμε να έχουμε εθελοντές αστυνόμους, όπως ακούω, ελπίζω να μην είναι αλήθεια. Ακούω ότι είναι στην Ιταλία που καταδίδουν τους μετανάστες και μετά τους βάζουν φυλακή. Τέτοιον εθελοντισμό εμείς δεν τον θέλουμε. Δεν θέλουμε έναν εθελοντισμό ο οποίος να δίνει τη δυνατότητα στα κράτη να μην ανταποκρίνονται στοιχειοδός σε υποχρεώσεις που έχουν. Ας πούμε στην Ελλάδα μας λείπουν 8.000 πυροσβέστες γι' αυτό το λόγο και γι' αυτό το λόγο γίναν πολλές πυρκαγιές που γίνανε έχουμε 120.000 εθελοντές πυροσβέστες εάν το κράτος δεν πάρει μέτρα δεν μπορούν 120.000 να λύσουν το πρόβλημα. Και πάει λέγοντας. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι εάν δεν αλλάξουν συνολικά κοινωνικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν τα προβλήματα της νεολαίας και των εργαζομένων δεν βρεθούν πραγματικά στο επίκεντρο των πολιτικών και των αναγκών, όσο εθελοντισμό και να κάνουμε, δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Και ο Στυλιάνοφ τελευταίος, στο Γιάννοφ συγγνώμη, μετά από, ναι, ο τελευταίος. Θα ήθελα ως... Ως ε, ε, κάποιος ο οποίος ε, έχω ασχοληθεί πολύ με τον εθελοντισμό. Και βέβαια το να είμαι μέλος του κόμματός μου ε, το κάνω εθελοντικά πράγματι. Είμαι και εθελοντικά πάλι μέλος μιας οργάνωσης ε, μη ε, κρατικής. Βεβαίω είναι εθελοντικά και αυτά. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προωθήσουμε την προσπάθεια του εθελοντισμού. Συμφωνώ με την προηγούμενη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον εθελοντισμό και πρέπει να ενθαρρύνουμε την εθελοντική δραστηριοποίηση των πολιτών. Δυστυχώς στη Βουλγαρία δεν έχουμε ε, ιδιαίτερο νόμο που να ρυθμίζει τα του εθελοντισμού. Στην ε, προηγούμενη Βουλγαρική Βουλή, όταν ήμουν ακόμη βουλευτής δηλαδή ε, στην Εθνική μας Βουλή, ανέλαβα την πρωτοβουλία να συντάξω ε, σχέδιο νόμου για να ρυθμιστούν τα, των εθελοντών και όλα τα σχετικά σε σχέση και με τη δημόσια τάξη και με το πυροσβεστικό σώμα με την αντιμετώπιση ατυχημάτων. Αυτό δε, το νομοσχέδιο εν τέλει απορρίφθηκε από τους σοσιαλιστές που είχαν τότε την πλειοψηφία στην Βουλγαρική Βουλή. Και εμένα αυτό με κατέπληξε, διότι εν τέλει πρόκειται για κοινωνικό έργο. Τώρα στη Βουλγαρία δεν έχουμε παρά μόνο μία πραγματικά εθελοντική οργάνωση και ε, ε, αυτή είναι ο βουλγαρικός ερυθρός σταυρός. Είναι πραγματικά δηλαδή εθελοντές οι άνθρωποι που ασχολούνται εκεί. Το να ε, κάνουμε το έτος 2011 έτος εθελοντισμού νομίζω πράγματι θα έχει μια θετική απήχηση και πιστεύω ότι θα συμβάλλει σε μια ενθάρρυνση και της νέας Βουλγαρικής Βουλής να ε, ρυθμίσει νομοθετικά το έργο των εθελοντών. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ντέλη, θέλετε να σχολιάσετε εν τέλει, η ψηφοφορία γίνεται αύριο, ε, ίσως δεν το ξέρετε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για όσα είπατε. Για μένα είναι φανερό ότι η εθελοντική δραστηριότητα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κοινωνική πολιτική, δεν έχει σαν ρόλο την υποκατάσταση αυτή, γιατί αυτό που είπατε για την εθελοντική αστυνομία ας πούμε. Αυτό το λέω όμως ρητά, ελπίζω να μην ε, έχω δημιουργήσει παρεξήγηση. Επίσης κάτι που μου φαίνεται σημαντικό αφορά την κοινωνική προστασία και ιδιαίτερα την υγεία. Έχουν ακουστεί πολλά ότι δηλαδή πολλοί εθελοντές δουλεύουν σε, για πια για την αποαμιαντοποίηση και εκτίθενται στον αμίαντο και αρρωσταίνουν. Πρέπει αυτό το έτος εθελοντισμού να επιτρέψει σε νέους και λιγότερο νέους να έχουν περισσότερη πρόσβαση στην κοινωνική περίθαλψη και η δική μας επιτροπή πρέπει να το κάνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άρα μπορεί να λήξει εδώ η συζήτηση για το έτος εθελοντισμού. Θα ψηφίσουμε αύριο σας υπενθυμίζω. Και τώρα περνάμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξής μας με τη συμμετοχή του Γενικού Υποδιευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης για την Περιφερειακή Πολιτική. Παρακαλώ να έρθουν εδώ οι αρμόδιοι στο Προεδρείο θα ακούσουμε την παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων της post αξιολόγησης των προγραμμάτων συνοχής. Καλωσορίζω την υποδιευθύντρια Κατερίνα Ματέρνοβα. Το 2007 η Κομισιόν και η Γενική της Διεύθυνση για την Περιφερειακή Πολιτική είχε αρχίσει αυτήν την εκ των υστέρων αξιολόγηση της περίοδου 2000 με 2006 και η τελική συνθετική αυτή αξιολόγηση θα τελειώσει τον Μάρτιο του 2010. Θα γίνει τότε η πλήρης παρουσίαση αλλά ήδη από σήμερα ζητήσαμε από εκπροσώπους της Γενικής αυτής Διεύθυνσης να μας παρουσιάσουν τα πρώτα αποτελέσματα ώστε από τώρα μέχρι το Μάρτιο όσοι και όσες ενδιαφέρονται να γνωρίζουν κάπως καλύτερα τι αντιπροσωπεύει η αξιολόγηση αυτή και να γίνει πιο εύκολα η πλήρης ακρόαση το Μάρτιο. Έχει αμέσως το λόγο η υποδιευθύντρια Ματέρνο. Ευχαριστώ Ντανούτα. Ακόμα και να μπορώ να μιλήσω σλοβακικά, θα συνεχίσω στα αγγλικά. Καλησπέρα σας λοιπόν. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ για να σας παρουσιάσω λίγο τόσο τη μεθοδολογία όσο και τα όσα κάναμε και κάποια από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν για την εκ των υστέρων αξιολόγηση για τους, ε, τα προγράμματα του 2000-2006 για την πολιτική συνοχή. Η κυρία Χούμπνερ είχε δίκιο όταν μίλησε για τις προκλήσεις της αξιολόγησης, διότι πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος παρουσιάζει πραγματικά επιπλοκές για μας και να σας αναφέρω για ποιους δύο-τρεις λόγους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει ασχοληθεί σε αρκετούς τομείς και για την πολιτική συνοχή, αλλά όχι μόνο για την πολιτική συνοχή και έχει λάβει επικρίσεις ε, γιατί δεν κάνει ίσως αρκετά καλές ε, αξιολογήσεις είτε εκ των προτέρων είτε εκ των υστέρων. Ε, μας χτύπησαν αυτές οι επικρίσεις τα τελευταία χρόνια, κυρίως το 2007 και προσπαθούσαμε να δούμε τα πράγματα ε, λίγο λιγότερο γραφειοκρατικά και να εξετάσουμε τα προγράμματα και τα έργα τα οποία είναι εξελίξη ε, και να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε τις αξιολογήσεις αυτές κατά τρόπον ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του τι γίνεται με την ε, πολιτική συνοχής διότι όλοι αγαπούμε και πιστεύουμε την πολιτική αυτή, αλλά ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να έχουμε τα δεδομένα τα οποία θα υποστηρίξουν ε, τους ισχυρισμούς για το κατά πόσον είναι καλή και αποτελεσματική η πολιτική μας. Ναι, ναι, ναι. Χρειαζόμαστε την προηγούμενη διαφάνεια. Να δούμε λίγο, λοιπόν, τι ακριβώς πρέπει να κάνει μια ομάδα αξιολόγησης. Έχουμε περίπου 230 προγράμματα ε, τα οποία ε, είναι σε μία κτίνα από 6 εκατομμύρια ε, προγράμματα των 6 εκατομμυρίων και μέχρι προγράμματα των 6 δισεκατομμυρίων. Έχουμε διάφορα διάφορες μορφές προγραμμάτων, διάφορες κυβερνητικέ διομές που εξετάζονται και για την Κομισιόν δύο ακόμα στοιχεία περιπλέκουν το θέμα της αξιολόγησης. Καταρχήν είναι η Κομισιόν αυτή η οποία είναι αρμόδια για την εκ των υστέρων αξιολόγηση και όχι τα κράτη-μέλη και στην πράξη ελάχιστα είναι τα κράτη-μέλη που κάνουν αξιολόγηση. Και επίση υπάρχει το θέμα της διάθεση των δεδομένων διότι η Κομισιόν είναι δύο στάδια μετά το όσα συμβαίνει, τα όσα συμβαίνουν επί τόπου. Για τα δεδομένα δεν υπάρχουν ε, ε, συμφωνημένοι και κωδικοποιημένοι δείκτες ε, για την αξιολόγηση, κυρίως για την αξιολόγηση την διασυνοριακή και αυτό είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Ναι. Επίσης, η αξιολόγηση έχει και ένα διτό στόχο ε, και να δούμε το ποιος είναι υπόλογος τι, αλλά και να μάθουμε και κυρίως το ποιος είναι υπόλογος γιατί ε, είναι ε, ο προεξάρχων λόγων. Προσπαθούμε να έχουμε κάποιες καινοτόμες προσεγγίσεις για να δούμε πώς μπορούμε να το υπερκεράσουμε το πρόβλημα αυτό. Τι κάναμε λοιπόν για την αξιολόγηση αυτή εξετάζοντας το διάστημα 2000-2006 στη Γενική Διεύθυνση Ρίτζο. Κάναμε μία κατανομή και απομακρυνθήκαμε από την προηγούμενη προσέγγιση που κάναμε μια συλλογική ε, αξιολόγηση όλων των προγραμμάτων και εξετάζαμε το σύμπαν ουσιαστικά και προσπαθούσαμε να κάνουμε μια αξιολόγηση αναστόχους, ε, να κάνουμε μια κατανομή των πακέτων και κάναμε μια αξιολόγηση σε 14 διαφορετικά πακέτα εργασίας ή 14 διαφορετικά προγράμματα. Αυτά που θα δείτε σήμερα ε, και για να, σας, ε, ε, να μην σας προκαταβάλω, δεν έχουμε την πλήρη αξιολόγηση έτοιμη ακόμα. Θα λαμβάνουμε αποτελέσματα από τώρα μέχρι το Μάρτιο του 2010 και αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι τα πρώτα τέσσερα σημεία, θα σας τα αναφέρει η Βορώνικα σε λίγο. Και αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να περάσουμε από τις ε, σχετικά μικρές ε, θεματοκές αξιολογήσεις, η πολιτική συνοχής και η ανάπτυξη της υπαίθρου, η διάσταση του φύλου, ε, στις πιο μεγάλες, εξετάζοντας τους μεγαλύτερους, τους συνολικούς στόχους και τις διάφορες θεματικές ενότητες αναμέσω, εξετάζοντας το κόστος ανα μονάδα για τα μεγαλύτερα προγράμματα και το πρώτο το οποίο θα αναφέρουμε είναι μια συνολική αξιολόγηση της διαχείρισης και, της, ε, και του συστήματος εφαρμογής. Όχι τον έλεγχο, αλλά το σύστημα διαχείρισης και εφαρμογής. Προσπαθήσαμε λοιπόν να ξεφύγουμε από τη συνολική εικόνα και να έχουμε ε, μία προσέγγιση σε μικρότερα πακέτα για να έχουμε μία συνολική εικόνα και να δημιουργήσουμε τελικά ένα μοσαϊκό του τι ακριβώς κάνει η πολιτική ε, συνοχή στους διάφορους τομείς. Σίγουρα δεν είναι τέλεια, σαφώς ε, χρήζει βελτιώσεων, αλλά ε, διαπιστώνουμε ήδη ότι είναι λίγο πιο δομημένα τα πράγματα και έχουμε λίγο πιο καλά αποτελέσματα από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Όλα αυτά τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στο ιστοσελίδα μας και οργανώνονται και διασκέψεις και εργαστήρια και ακροάσεις με όσους κάνουν την αξιολόγηση, με ομοτήμους, με ακαδημαϊκούς και προσπαθούμε επίσης να δούμε λίγο και την ε, μεθοδολογία και προσπαθούμε να κάνουμε και κάτι καλύτερο για το μέλλον. Εδώ να αναφέρω και τη διάσκεψη που θα γίνει στο τέλος του μηνός ε, στη Βαρσοβία. Ε, θα είναι ο Επίτροπος Αμίτς και εκεί, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ε, θα γίνει μια διάσκεψη λοιπόν για τις μεθοδολογίες αξιολόγησης για το μέλλον. Θα υπάρχουν άτομα τα οποία κάνουν αξιολογήσεις από όλα τα κράτη-μέλη ε, καθώς και ακαδημαϊκοί και άτομα από άλλους διεθνούς οργανισμούς που ασχολούνται με αντίστοιχα προβλήματα για να προσπαθήσουμε λίγο να κάνουμε μια βολιδοσκόπηση, μια ανταλλαγή απόψεων για το πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα στο μέλλον. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι βανάγνωστο αυτό που βλέπετε, αλλά είναι για να έχετε μία εικόνα. Έχετε όλη τη διαφάνεια από ό,τι άκουσα, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχω προβλήματα, δεν έχω τα γυαλιά μου, μάλλον θα γυρίσω στην οθόνη λοιπόν. Βλέπετε εδώ Έχουμε τα 14 πακέτα τα οποία είναι χωρισμένα σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες. Έχουμε τα συστήματα διαχείρισης και εφαρμογής. Αυτό είναι αυτό για το οποίο έχουμε αποτελέσματα ήδη σήμερα να σας παρουσιάσουμε. Έχουμε το δεύτερο που είναι ε, το μπλοκ των δεδομένων, το πώς συλλέγονται τα δεδομένα και το κόστος αναμονάδα σε μεγάλα προγράμματα. Και αυτό το έχουμε εδώ σήμερα. Μετά έχουμε το θεματικό μπλοκ, την υποστήριξη από τις επιχειρήσεις, ε, αλλαγές στο περιβάλλον και στο κλίμα, μεταφορές, ε, ε, διαρθρωτικές αλλαγές και παγκοσμιοποίηση, η διάσταση του φύλου και τα δημογραφικά θέματα και η ανάπτυξη της υπαίθρου. Τα δύο τελευταία τα έχουμε, θα σας τα αναφέρει Βερόνικα σε λίγο και τέλος έχουμε ένα μπλοκ με μοντέλα τα οποία χρησιμοποιήσαμε, ε, μακροοικονομικά μοντέλα για την ε, ε, πολιτική έχουμε το Hermin, το Quest και το Trans Tools. Διστάσαμε λίγο να σας δώσουμε αυτή τη διαφάνεια Βέβαια τα έχετε σε αντίγραφα και που σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερο ο δισταγμά μα. Ε, ε, τα μηνύματα δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να τα βάλουμε γιατί είναι λίγο πρόημο αυτή τη στιγμή να συζητάμε για μηνύματα. Οι εξολογήσει είναι εν εξελίξει και θα χρειαστούμε λίγο ακόμα χρόνο για να έχουμε μια συνολική εικόνα, ένα συνολικό μήνυμα. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι έχουν επιτευχθεί αρκετά καλά πράγματα με τι πολιτικέ του παρελθόντο, αλλά υπάρχουν κάποιε δομικέ διαφορέ. Μία εξ αυτών είναι έλλειψη στρατηγικού ε, προσανατολισμού σε κάποιου τομεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε. Καλύτερη κατανομή πόρων και να εστιάσουμε λίγο καλύτερα στα αποτελέσματα. Και πάλι όμω. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε την προηγούμενη διαφάνεια. Στην κάτω αριστερά γωνία ε, του θεματικού μπλοκ νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη και πιο δομημένη εικόνα στα αποτελέσματα. Γι' αυτό ακριβώς ελπίζουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από την αξιολόγηση όσο προχωρά ο χρόνος. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ με την εισαγωγή μου. Η Βερόνικα θα σας παρουσιάσει τις τέσσερις αξιολογήσεις που έχουμε ήδη κάνει και από εκεί και πέρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε πρώτα στην αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης και εφαρμογής. Ε, δεν εξετάζουμε το θέμα της εποπτείας, αλλά των συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για να εφαρμοστεί η πολιτική συνοχής. Η μελέτη αυτή έγινε από το EPRC, στο Strathclyde, στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde στη Γλασκόβη και ε, ο επικεφαλής ήταν ο καθηγητής Τζον Μπάχτλερ με ε, μια αυστριακή εταιρεία συμβούλων Είχαμε μια κοινοπραξία, είχαμε 50 άτομα τα οποία ασχολήθηκαν με αυτή την αξιολόγηση για να δουν τα συστήματα εφαρμογής για την πολιτική συνοχής. Είδαμε σχεδιασμό προγραμμάτων, επιλογή προγραμμάτων, ε, χρηματοδότηση ε, και εταιρικέ σχέσεις. Και από τα 14 πακέτα της αξιολόγησης, αυτό είναι αυτό το οποίο εστίασα περισσότερο στις 10 ε, νέες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι θεωρήσαμε ότι θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσουμε πόσο καλά τα κράτη-μέλη τα οποία εντέχθηκαν το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δημιουργήσει συστήματα για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος όγκος ε, πληροφοριών για αυτή την αξιολόγηση, τα οποία δημοσιεύεται όλο στην ιστοσελίδα μας, επομένως αν σας ενδιαφέρει μπορείτε κάλλιστα να την επισκεφτείτε. Στην αξιολόγηση τώρα ε, λαμβάνουμε υπόψη και εθνικές εκθέσεις. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές εκθέσεις για τα συστήματα διαχείρισης και εφαρμογής για τις 10 νέες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν και σημαντικά αποτελέσματα από την αξιολόγηση για τις χώρες αυτές. Το βασικό μου συμπέρασμα είναι ε, καταρχήν ε, ότι δημιουργήθηκαν συστήματα για τις νέες χώρες για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής το διάστημα 2004-2006 Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό επίτευγμα από μόνο του. Και το άλλο το οποίο διαπιστώνεται κατά την αξιολόγηση είναι ότι μπορεί τα προγράμματα να ήταν πολύ περίπλοκα και να υπήρχε μεγάλη γραφειοκρατία αρχικά. Τα συστήματα τελικά εξορθολογίστηκαν και ήταν πιο αποτελεσματικά συν το χρόνο. Το άλλο σημείο είναι ότι ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν και θετικά στοιχεία από τα εσωτερικά ε, συστήματα διαχείρισης. Η Πολωνία είναι ένα καλό παράδειγμα όπου τα συστήματα πολιτικής συνοχής άρχισαν να μεταφέρονται και στις εσωτερικές τους πολιτικές. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης και για τις, χώρες, τις νέες χώρες ένταξης και για τις 15 ε, παλαιότερες χώρες είναι ότι υπάρχει μια ανάγκη να αυξηθεί η στρατηγική διαχείριση να αυξήσουμε λοιπόν τα, ε, τη στρατηγική μας, ε, το στρατηγικό μας προσανατολισμό στο τι επιτυγχάνεται και στο πώς δαπανούνται σωστά τα κονδύλια. Ναι, μεν είναι σημαντικό και αυτό, αλλά θα πρέπει να εστιάζουμε κυρίως και στα αποτελέσματα. Οι συστάσεις που γίνονται στην αξιολόγηση ε, εστιάζουν πάρα πολύ σε αυτό το θέμα των αποτελεσμάτων της πολιτικής ε, και στο να παρουσιάζονται αυτά περισσότερο το γεγονός επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο και να προάγει τις ε, δυνατότητές τους, διότι τα συστήματα τα οποία προκύπτουν ε, για τα συστήματα διαχείρισης ε, είναι πολύ σημαντικό να είναι τα βασικά και επίσης έχουμε μεγαλύτερη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Αν κάποια κράτη-μέλη λοιπόν έχουν αναπτύξει κάποιε καλέ ε, πολιτικέ διαχείριση, καλό θα ήταν να τι γνωρίζουν τα άλλα κράτη-μέλη και να μπορούν να μάθουν ο ένα από τον άλλον. Αυτή τη στιγμή λοιπόν συζητάμε τα ευρήματα αυτής της αξιολόγησης και τι ακριβώς θα αποφασίσουμε για το μέλλον της πολιτικής. Θέλουμε να επανεξετάσουμε κάποια από τα όσα διαπιστώσαμε όταν θα έχουμε και τα στοιχεία από τις υπόλοιπες αξιολογήσεις, ώστε όταν θα έχουμε τα συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής, να επανεξετάσουμε και τα θέματα της αποτελεσματικότητας εφαρμογής διότι δεν θέλουμε να έχουμε τέλεια ε, συστήματα εφαρμογής αν δεν έχουμε αποτελεσματικές πολιτικές. Θέλουμε αυτά τα δύο να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Έχουμε πολύ υλικό λοιπόν για τα συστήματα αυτά. Να περάσω τώρα σε μία πολύ μικρότερη ε, μελέτη ε, για το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα θέματα φύλου και τα δημογραφικά θέματα. θεωρούμε βέβαια ότι αυτά τα θέματα είναι πιο σχετικά για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά θέλαμε να δούμε τι γίνεται με το θέμα του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα θέματα αυτά. Ε, μία Ιταλική κοινοπραξία εξέτασε τα θέματα, η NUS και CISIL και καταλήξανε και στο συμπέρασμα ότι και τα δύο αυτά ε, θέματα είναι σημαντικά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά υπάρχουν διαφορές μεταξύ των. Για τα δημογραφικά θέματα, αυτά δεν ήταν προτεραιότητα το 2000 όταν αναπτύχθηκαν αυτά τα προγράμματα. Ωστόσο, η αξιολόγηση διαπιστώνει ότι ε, έχουν υποστηριχθεί προγράμματα ε, για να ε, βοηθήσουμε περιφέρειες που ασχολούνται με τις δημογραφικές αλλαγές. Όσον αφορά το θέμα του φύλου, το φύλο ήταν μια οριζόντια προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης το 2000 και υπάρχουν πολλά στα προγράμματα που αφορούν στις συνιστώσεις του φύλου. η αξιολόγηση βέβαια καταλήγει στο συμπέρασμα ήταν ότι είχαμε περισσότερα λόγια παρά πράξεις τα σχετικά προγράμματα υποστηρίχτηκαν, υπάρχουν και παραδείγματα στην αξιολόγηση, αλλά πολλές φορές ε, το θέμα του φύλου ήταν ε, το θέμα της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις και δεν προσπαθήσαμε να επιτύχουμε κάτι για το ίδιο το θέμα ουσιαστικά. Στις συστάσεις ε, λέμε ότι τα θέματα του φύλου και τα δημογραφικά θέματα θα πρέπει να είναι προτεραιότητες όπου υπάρχει σχέση για τις περιφέρειες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το άλλο στοιχείο το οποίο προκύπτει από την αξιολόγηση είναι ότι το τοπικό επίπεδο είναι σημαντικό. Ε, θα πρέπει να υπάρχει εθνική νομοθεσία για να ασχολείται με θέματα φύλου και δημογραφικά θέματα αλλά ε, σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν στρατηγικές οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις ε, στα θέματα αυτά. Εμείς ε, στην Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο θεωρούμε ότι θα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο τις οριζόντιες προτεραιότητες στο μέλλον, διότι εάν υπάρχουν πάρα πολλές οριζόντιες προτεραιότητες μπορεί να μην έχουμε ουσιαστικές προτεραιότητες. Το θέμα λοιπόν είναι εάν υπάρχει ένας κατάλογος οριζόντιων προτεραιοτήτων ίσως θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις περιφέρειες να σκεφτούν ποιες είναι οι πιο σημαντικές για αυτούς και όχι να προσπαθήσουν να έχουν προσκελέστα το κατάλογο 12 π.χ. προτεραιοτήτων που θα πρέπει να σέβεται ο καθένας. Η επόμενη αξιολόγηση που θα αναφέρω είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ανάπτυξη τη Υπαίθρου. Αυτή ήταν η μικρότερη από τι μελέτε αξιολόγηση. Ήταν σε πειραματικό στάδιο. Ε, εξετάσαμε μόνο πέντε κράτη-μέλη και προσπαθήσαμε να δούμε ποιο είναι ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερική Ανάπτυξη για την ανάπτυξη πέθρου σε αυτά τα κράτη-μέλη. Η μελέτη έγινε από μια αυστριακή εταιρεία συμβούλων, τη ΜΕΤΙΣ, και το πρώτο θέμα το οποίο χρειάστηκε να ασχοληθεί ήταν ότι δεν υπάρχουν απλοί ορισμοί ούτε για τις περιοχές της υπαίθρου, ούτε για την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτό ήταν η πρώτη πρόκληση λοιπόν για την αξιολόγηση και η πρόκληση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη διότι η ανάπτυξη της υπαίθρου πολλές φορές ορίζεται με τελείως διαφορετικό τρόπο σε κάθε κράτος μέλος και αυτό που θεωρείται ύπεθρος για ένα κράτος μέλος μπορεί να μην θεωρείται ύπεθρος για ένα άλλο και υπάρχουν πολλές <laughs> ε, πολιτισμικές, ιστορικές ε, διαφορές οι οποίες δημιουργούν διαφορετική αντίληψη για το ποια περιοχή θεωρείται περιοχή της υπαίθρου ή όχι για την ανάπτυξη της υπαίθρου τώρα και πάλι δεν υπάρχει μία θεωρία για την ανάπτυξη της υπαίθρου ε, και ε, προκύπτουν συμπεράσματα από διάφορες οικονομικές θεωρίες. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, συνεισφέρει σημαντικά στις περιοχές της υπαίθρου και στις χώρες που εξετάσαμε είχαμε περίπου 25% της χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις περιοχές της υπαίθρου. Αλλά οι περιοχές, οι εν λόγω περιοχές δεν θεωρούσαν ότι θα δαπανούνται τόσο μεγάλα κονδύλια για αυτούς. Ε, εξετάσαμε στις ασθενέστερες περιοχές, είτε είναι αστικές είτε είναι περιοχές της υπαίθρου και θεωρούμε ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση και αυτό το οποίο προκύπτει από την αξιολόγηση είναι ότι η ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο είναι σημαντική και θα μπορούσαν ίσως μηχανισμοί τοπικής ανάπτυξης να ενισχύσουν ε, την ε, σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου της ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον τρόπο με τον οποίο το αντιλαμβανόμαστε. Η τελευταία μελέτη για την οποία θα σας ε, παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία ε, είδε το κόστος αναμονάδα των μεγάλων προγραμμάτων. Είναι λίγο διαφορετικό αυτό και όπως είπε και η Καταρίνα απλά σας δίνουμε εικόνες από τελείως διαφορετικές οπτικές γωνίες της ε, πολιτικής. Ελπίζουμε στο τέλος στην τελική έκθεση να τα συγκεράσουμε όλα μαζί. Εδώ είχαμε μεγάλα προγράμματα προγράμματα υποδομών ε, άνω των 50 εκατομμύριων ευρώ τα οποία αποφασίστηκαν ξεχωριστά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπήρχε και ανάγκη να γίνει και ανάλυση κινδύνου για τα προγράμματα αυτά. Εμείς ως Γενική Διεύθυνση Ρίτζο θέλαμε να δούμε αν μπορούμε να εξετάσουμε ε, πιο διεξοδικά το κόστος αναμονάδα σε, αυτές, σε αυτά τα προγράμματα. Την μελέτη την ανέλαβε μια κοινοπραξία που περιλαμβάνει την RGL, τη Forensic Accounts, τη Frontier Economics και μία ακόμα εταιρεία και είχαμε λοιπόν συμβούλους οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι ακριβώς κάνουν και μπορούσαν να δουν μεγάλα προγράμματα υποδομών. Η μελέτη ήταν προγράμματα και πάλι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ε, θα αναπτύξουμε ε, το θέμα του Ταμείου Συνοχής και του ΙΣΠΑ αργότερα. Ε, η μελέτη διαπίστωσε ότι πολλά από τα προγράμματα υπερέβησαν τον προπολογισμό τους, ε, αλλά πολλά τήρησαν το στόχο τους. 75% των προγραμμάτων καθυστέρησαν. Αυτό βέβαια δεν μας ανησυχεί πολύ, γιατί αυτό συνάδει με τους διεθνείς κανόνες. Δεν είμαστε καλύτεροι λοιπόν από ό,τι γίνεται διεθνώς, αλλά δεν είμαστε και χειρότεροι. Η αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη να εστιάσουμε περισσότερο στην ανάλυση κινδύνου και στον μετριασμό των κινδύνων σε αυτά τα μεγάλα προγράμματα και γίνονται και κάποιες συστάσεις προς εμάς για το πώς μπορούμε να το κάνουμε και το πώς θα μπορούσε να είναι κοινή η κατανομή του κινδύνου μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το τι γίνεται με τα προγράμματα. Ένα από τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέραν ιδιαίτερα στη μελέτη αυτή είναι κατά πόσον είναι εφικτό και δυνατό να έχουμε μία βάση δεδομένων του κόστου αναμονάδα των μεγάλων ε, προγραμμάτων υποδομών ώστε να έχουμε benchmark ε, και σημεία αναφοράς για προγράμματα πολιτικής συνοχής. Το σκεπτικό δεν είναι να πούμε ότι όλα τα προγράμματα αυτοκινητοδρόμων έχουν ένα συγκεκριμένο κόστος, αλλά να μπορούμε να κάνουμε μία σύγκριση αναλόγων προγραμμάτων, να δούμε τι κόστος υπήρχε σε κάθε περίπτωση και τα κράτη-μέλη να βοηθούν άλλα κράτη-μέλη με τα δικά του προγράμματα και την εφαρμογή τους. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι δυνατόν και επίσης ε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν βάσεις δεδομένων και αυτό είναι ένα κενό το οποίο θα μπορούσε να πληρώσει η Γενική Διεύθυνση Ρέτζου. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε και να υπάρχει κάποιο όσφελος, ε, να βοηθήσουμε και τα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη μεγάλων προγραμμάτων. Συζητάμε ε, με την ERB για να δούμε αν μπορούμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και να προχωρήσουμε το θέμα αυτό. Θα τα αναπτύξουμε αυτά περαιτέρω στην ε, αξιολόγηση του Ταμείου Συνοχής και της ΙΣΠΑ που θα αρχίσει στις αρχέ του επομένου έτους και θα συνεχίσει μέχρι το 2011. Αυτά λοιπόν ως μια μικρή ε, φωτογραφία των ε, τεσσάρων στοιχείων ε, που έχουμε από, τα από τις 14 θεματικές ονότητες που εξετάσαμε και όπως είπε και η Κατερίνα θα είμαστε στη διάθεσή σας για νέα στοιχεία όταν θα τα έχουμε και εμείς στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ. Για την παρουσίασή σας. Τώρα επιθυμείτε να ρωτήσετε να σχολιάσετε. Δεν είναι απαραίτητο να ληφθεί απόφαση σήμερα. Πρόκειται περισσότερο για να διευρύνεται την κατανόηση των διαστάσεων της πολιτικής συνοχής. Ποιος να το λεπτό, εσείς κύριε. Α, όχι, η κυρία Μπίαρντερ. Είναι πολύ ενδιαφέρον να επανέρχεται κανείς στην έρευνα ε, των ε, διαφόρων project όπου ήδη γνωρίζετε πώς έχουν προχωρήσει, αλλά βλέπετε έτσι τις ρίζες. Όταν είπατε για τις προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων και για τα δημογραφικά που θεωρήσατε ότι ε, δεν είναι αρκετά. Το κατανοώ αυτό. Αλλά να μην αφαιρεθούν όμως οι προτεραιότητες διότι αποκτήθηκαν με αγώνα ώστε να υπάρχουν αυτές οι checklist όταν δίνονται τα κονδύλια να ε, ισχύουν αυτές οι προτεραιότητες. Ε, να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αυτές οι καλές κοινωνικές προτεραιότητες και να αναγνωρίζονται, να τους αποδίδεται η αναγνώριση που τους αξίζει. Όπως είπα, κατακτήθηκαν μετά από πολλούς αγώνες και πολλά χρόνια. Και δεν θα ήθελα να διαβρωθούν. Δεν έχει μικρόφωνο, ο κ. Ε, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρωτοβουλία και να συγχαρώ τις ε, δύο κυρίες για την ε, παρουσία που κάνανε. εμένα με εντυπωσίασε, με εντυπωσίασε θετικά θα θέλω να πω και ελπίζω και στο μέλλον να έχουμε παρόμοιες. θα ήθελα να θέσω τρεις ερωτήσεις, αν μου επιτρέπουν η, κυρία Πρόεδρος οι κυρίες... Ε, είναι απλές, δεν είναι δύσκολες. Η πρώτη ερώτηση αφορά τις πέντε χώρες για τις οποίες έγινε έρευνα ε, του Ταμείου Συνοχής και είχαν και ύπεθρο και αγροτικές ε, περιοχές. Ποιες είναι αυτές οι πέντε χώρες, αν μπορούν οι κυρίες εισηγήτριες να μας πούν. Η δεύτερη ερώτηση που έχω να κάνω είναι στο κριτήριο της υπαίθρου. Σωστό είναι αυτό ότι είναι δύσκολο να προσδιορίσει από χώρα σε χώρα τι είναι ύπεθρος. Ε, στη μελέτη που έγινε πάρθηκε υπόψη το ποσοστό αγροτικής παραγωγής στην περιοχή της ύπεθρου ή αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν έγινε ακατανοητός εάν η αγροτική παραγωγή εγινα κατανοητο εαν η κριτήριο για να πούμε ότι μια περιοχή είναι ύπεθρος ή όχι ή και πόσο ψηλό είναι αυτό το ποσοστό εν πάση περιπτώσει. Και μια τελευταία ερώτηση ε, έχει να κάνει με το ποια είναι η γνώμη της ερευνητικής ομάδας για το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ή αν πρέπει να υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο αντίστοιχες μονάδες ε, μελέτης των αποτελεσμάτων της ε, πολιτικής συνοχής. Δηλαδή νομίζω ότι είναι, θα ήταν πολύ σημαντικό αν σε κάθε χώρα μέλους της Ένωσης υπήρχε μια αντίστοιχη μελέτη για το σύνολο των προγραμμάτων, ώστε και οι πολίτες των χωρών μελών να ενημερώνονται πιο γρήγορα και πιο άμεσα. Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, αλλά δεν θέλω να πάρω το χρόνο σας. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Με ενδιαφέρει πρώτα εάν θα μας δοθούν οι μελέτες αυτές κατόπιν ετησιός μας. Η αξιολόγηση με ενδιαφέρει πολύ. Το θέμα για την ισότητα των φύλων και το λεγόμενο mainstreaming που ήταν Μέγα αγώνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2000 και έχουμε επιτύχει και βελτιώσεις. Έχουμε και εμεί κάνει μια μελέτη που κατέληξε στα ίδια συμπεράσματα με εσά, ότι δηλαδή όντως υπάρχει διαφορά εάν δοθούν τα χρήματα δηλαδή ειδικά για ένα φύλλο ή εάν άντρες και γυναίκες μπαίνουν στο ίδιο καλάθι και οι γυναίκες που ε, ιδρύουν επιχειρήσεις δεν ε, έχουν ευκαιρίες διότι δεν ενθαρρύνονται, δεν προωθούνται συγκεκριμένα. Το ίδιο διότι οι γυναίκες συχνά έχουν διαφορετικές ανάγκες από τους άντρες ε, ανατομέα. Έχει λοιπόν διαφορά και επίσης εάν η συλλογή στατιστικών δεδομένων γίνεται αναφύλο Για να καταλήξουμε σε αυτά τα συμπεράσματα πέρασε και χρόνος. Τώρα, εγώ δεν είμαι συμφωνή με ένα συμπέρασμα που λέτε δηλαδή ότι, ότι αυτή η γενική αρχή δεν λέω ότι πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο αλλά είναι μια βασική αρχή ότι λέει, λέτε δεν είναι απαραίτητο. Πρώτον, περιλαμβάνεται στη συνθήκη. Δεύτερο, είναι απαραίτητο, διότι και στην ε, περιοχή όπου προέρχομαι εγώ έχουμε κάνει αναλύσεις. Αυτές λένε μεν στη θεωρία ότι, έχουν, ότι έχει εκπληρωθεί το κριτήριο, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν ληφθεί υπόψη ιδιαίτερε ανάγκε των γυναικών. Γι' αυτό με ενδιαφέρει η μελέτη αυτή και το θέμα του κινδύνου, της ανάλυσης ωφέλους κινδύνου και αυτά έχουν συζητηθεί εδώ πολύ στο Κοινοβούλιο και διαμακρών. Και συχνά οι προτάσεις μας αγνοήθηκαν από την Επιτροπή και ούτε έχουν μελετηθεί αρκετά. Και η μελέτη σας αποδείχνει ότι το Κοινοβούλιο, δείχνει, ε, το κοινοβούλιο είχε δίκιο. Με ενδιαφέρουν λοιπόν και τα συμπεράσματα. Μπορείτε να μας τα διαθέσετε γραπτό στα συμπεράσματα που εξάγεται από τις μελέτες αυτές και γενικά τις μελέτες μπορούμε να τις έχουμε γραπτές. Νομίζω δεν είναι και η τελευταία φορά που θα τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα γιατί θα κληθούμε και στο μέλλον να αναζητήσουμε, να βρούμε μηχανισμούς, πώς μπορούμε δηλαδή και με λιγότερη γραφειοκρατία αλλά και με τη ρίση των αρχών και με περισσότερη συνέπεια να ε, διαθέτουμε τα ε, χρήματα των κονδυλίων. Ευχαριστώ. σε σχέση με την έρευνα για το management ακούμε από αυτούς που ηγούνται τον project ότι θέλουν και προτείνουν απλούστευση των διαδικασιών. Κατά πόσον έπαιξε το θέμα αυτό ένα ρόλο στη μελέτη σας. Και επίσης οι project manager, οι ε, κοινότητες, οι περιφέρειες ρωτήθηκαν σχετικά. Έγινε δηλαδή αυτή η διερεύνηση το, από την πλευρά των ενδιαφερομένων και ποιε βελτιώσει μπορεί να προκύψουν σύμφωνα με τις προτάσει τους. Μία ερώτηση ακόμα. Ο κύριο Τσέλερ. Μία... Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη μελέτη. Ω νέο Ευρωβουλευτή και επομένω είμαι στη φάση που μαθαίνω ακόμη, θέλω να επανέλθω σε μια συζήτηση που κάναμε στην αρχή της συνεδρίασής μας, όταν για μία ώρα και πλέον μιλήσαμε για ένα έγγραφο το οποίο δεν υπάρχει ακόμα ή εν πάση περιπτώσει είναι ένα έγγραφο πάντως το οποίο δεν έχουμε λάβει με επίσημο τρόπο και του οποίου ο αποστολέας είναι ακόμα ασαφές ποιος είναι και υποτίθεται ότι από το 2014 θα αρχίσει μια νέα στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα από τη μελέτη σας και από τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματά σας που και εμένα με ενδιαφέρουν πολύ και ελπίζω να συνεχίσουν οι μελέτες αυτές. Διαπιστώνω ότι η πολιτική συνοχής έχει πετύχει πολλά πράγματα, αλλά υπάρχουν και αδύναμα σημεία. Και στο στρατηγικό ε, θέμα και στρατηγική δηλαδή, αλλά και στους πόρους της. Αλλά και οι διάφορες παρεμβάσεις των συναδέλφων δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί πολλά project, αλλά δεν γνωρίζουμε καλά ποια είναι η αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής. Το θεωρώ αυτό που λέω και ως έκκληση για όλους μας και όλες μας εδώ στην Επιτροπή μας και επειδή η διαδικασία της Λισαβόνας θα αρχίσει τώρα πια να αποδίδει να δούμε αφενός πού καταλήγουν τα κονδύλια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιο αποτέλεσμα πετυχαίνουν. Επαναλαμβάνω, σας ευχαριστώ για τις μελέτες και ελπίζω να μας ε, διαβιβάσετε και τα αποτελέσματα. Ας απαντήσουν τώρα οι δύο κυρίες και μετά ε, συνεχίζουμε. Ευχαριστώ και για την αξιολόγηση που κάνατε ότι δεν είναι χαμένος χρόνος οι μελέτες αυτές. Πρόκειται για εκ των υστέρων αξιολόγηση της ε, περίοδου 2000 και 2006, επομένως ορώμενη εκ των υστέρων. Και γι' αυτό ο κύριος που ε, ρώτησε σχετικά με την απλοποίηση των κανόνων. Εγώ θα επανέλθω αύριο το πρωί και μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε για την απλοποίηση των κανόνων για την παρούσα περίοδο 2007 έως 2013. Για οτιδήποτε δηλαδή έχει σχέση με την περίοδο μετά το 2007. Διότι είναι ξεχωριστή η ρυθμιστική δομή της κάθε περίοδου σε ό,τι αφορά και τις ε, ρυθμίσεις ε, και Ελπίζουμε βέβαια αυτά που απέδωσαν οι μηχανισμοί που απέδωσαν καλά αποτελέσματα να μην ε, καταργηθούν για την επόμενη περίοδο και επειδή ε, το κάθε ένα γίνεται με ειδική ρύθμιση για κάθε χρηματοδοτική περίοδο αντιμετωπίζονται τα πλέον επίκαιρα θέματα μέσα σε αυτή την περίοδο. Μία από τις αρχές για την περίοδο 2007 έως 2013 ήταν η αυξημένη ανησυχία για το οικονομικό management. Και αυτό συζητούμε και στο Συμβούλιο τώρα και ελπίζουμε ότι και εσείς σύντομα θα το συζητήσετε εδώ στο Κοινοβούλιο. Πώς μπορούν λοιπόν να απλοποιηθούν ορισμένοι ε, κανόνες χωρίς να υπονομευθούν οι βασικοί πυλώνες της περίοδου αυτής. Τώρα, τούτη εδώ μελέτη είναι για την προηγούμενη περίοδο, για το παρελθόν επομένως. Και Ε, αναγνωρίζω την ανησυχία που εξέφασαν δύο κυρίες σχετικά με την ισότητα των φύλων. Υπάρχει μια συνολική ανησυχία σχετικά με ένα πληθωρισμό οριζόντιων, οριζόντιων προτεραιοτήτων που δεν αναφέρεται ειδικά στην προτεραιότητα για την ισότητα των φύλων. Συμφωνώ ότι ήταν μια ε, σκληρή μάχη που κερδίθηκε και ε, ότι πρέπει να διατηρήσουμε τις προτεραιότητες αυτές. Θα παραμείνουν αυτές οι προτεραιότητες. Ε, έχουμε σιγά σιγά όμως μια, ένα πληθωρισμό άλλων οριζόντιων προτεραιοτήτων. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, η ιδέα δηλαδή είναι να δώσουμε στις managing authorities το μέλλον τη δυνατότητα αφού ορισμένε προτεραιότητε, ορισμένε οριζόντιε προτεραιότητε θα παραμείνουν. Αλλά να μην βάζουν κάθε επίκαιρο θέμα ε, κάθε θέμα να μην μπαίνει δηλαδή ταυτόχρονα ε, ως ε, οριζόντια προτεραιότητα. Αυτή είναι η ανησυχία. Χωρίς όμως, όπως είπα, να ε, θέσουμε σε κίνδυνο την αρχή της ισότητας των φύλων, γιατί νομίζω ότι τα project μπορούν να είναι διαφορετικά και θα είναι διαφορετικά εφόσον ε, ενταχθεί ήδη στο προγραμματισμό τους το, η αρχή της ισότητας των φύλων. Τώρα, για την διαθεσιμότητα της. Βρίσκεται τις μελέτες αυτές ήδη στο διαδίκτυο. Θα βρείτε το, το σχετικό link στις παρουσιάσεις, στα φύλλα που σας δώσαμε δηλαδή, στην τελευταία σελίδα. Στη τελευταία, στο, στο τέλος της σελίδας αυτής θα βρείτε το, στη σελίδα 3. Α, στη σελίδα 3. Κάτω από εκεί που λέει καινοτόμε προσεγγίσεις, innovative approaches. Και ε, θέλουμε μάλιστα και πολύ να ε, ακούσουμε τις αντιδράσεις σας, γιατί ε, θα μας βοηθήσετε και στην τελευταία συνοπτική έκθεση που θα κάνουμε, αλλά θα βοηθήσετε και τους συμβούλους και μας να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει και τις αρμοδιότητες που μας δόθηκαν Δηλαδή θα μπορέσετε και να δείτε πόσο καλά ανταποκρίθηκαν οι ε, σύμβουλοι διαχείρισης. Τα βλέπετε λοιπόν όλα αυτά, τα έχετε διαθέσιμα όλα αυτά και μπορείτε να μπείτε στη συζήτηση. Σε ό,τι αφορά την διάσταση της υπαίθρου. Η συζήτηση για το τι είναι και τι είναι υπαίθρος διεξάγεται από καιρό. Αυτό που ισχύει τώρα είναι ο ορισμός του ΟΣΑ. Και αυτά η δουλειά που έγινε στην αξιολόγηση ήταν πάντοτε με βάση τον ορισμό του ΟΣΑ που εξετάζει με το κριτήριο της πυκνότητας του πληθυσμού. Αστικά κέντρα, ε, περιοχές υπαίθρου. Οι πέντε χώρες που επιλέχτηκαν ήταν η Γαλλία, η Γερμανία, Πολωνία, Σουηδία και Ισπανία. Και άλλη μια ερώτηση, ε, α, θα σας απαντήσει η Βερόνικα σε αυτήν. Εάν υπάρχουν παρόμοιες ε, μονάδες σε άλλες χώρες. Αυτές υπάρχει η κατανομή μεταξύ ε, κομισιών και χωρών μελών. Η Management authority είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση εκ των προτέρων. Τώρα, οι γίνονται αξιολογήσεις που πρέπει να γίνουν, τις κάνουν δηλαδή οι χώρες. Τώρα, ο κανονισμός δίνει ωστόσο στην Κομισιόν την αρμοδιότητα να κάνει την εκ των υστέρων αξιολόγηση. Εγώ θα προτιμούσα αυτό να μοιράζεται λιγάκι, να το μοιραζόμαστε λιγάκι με τις χώρες μέλη, ώστε δηλαδή να γίνεται πιο μοιρασμένα η προσπάθεια αξιολόγηση για τα αποτελέσματα. Ορισμένε χώρε μέλη το κάνουν, αν και δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα θέλαμε να συζητήσουμε για το μέλλον, δηλαδή να δώσουμε μια ενίσχυση σε αυτό το ρόλο των χωρών. Η Πρόεδρος, να προχωρήσουμε. Κυρία Ντέλη. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Στην μελέτη για την ανάπτυξη της υπαίθρου λάβατε υπόψη στις πέντε χώρες την πολιτική της ανάπτυξης των αστικών κέντρων γιατί υπάρχουν διασυνδέσεις ανάμεσα στην ανάπτυξη των αστικών κέντρων και της υπαίθρου. Η πολιτική, για παράδειγμα, των μεγάλων έργων υποδομής. Έχετε λάβει υπόψη το στοιχείο αυτό στη μελέτη σας. Όλμπριχτ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σχετικά με την δομή της αξιολόγησης εξ όσων κατανοώ η άντε, δηλαδή των προτέρων αξιολόγηση γίνεται την ώρα που ήδη τρέχει η επόμενη ε, περίοδος δηλαδή ε, προγραμματίζεται την επόμενη περίοδο χωρίς να ε, ε, είναι διαθέσιμη η περίοδος και μετά τα συμπεράσματα θα χρησιμοποιηθούν μετά από το 2014 ή θα χρησιμοποιηθούν μέσα στην περίοδο χρηματοδότησης, δηλαδή 2010 έως 2014. Δηλαδή εννοώ το εξής και έχει σχέση με την στρατηγική Ίσως ε, η διατύπωση να είναι διπλωματική, αλλά θα πω τι διαβάζω εδώ. Η μεγέθυνση των ε, συνεπειών δεν υπήρξε λόγο. Εγώ το βρίσκω αυτό διπλωματικό, δηλαδή διπλωματική διατύπωση. Αν καταλαβαίνω καλά, αυτό σημαίνει ότι εάν οι πόροι ήταν πιο ξεκάθαρα διατεθειμένοι για στρατηγικά θέματα που φαίνεται πως δεν είναι. Αν λοιπόν ήταν πιο ξεκάθαρα διατεθειμένη για αυτό το λόγο ή αν δεν ήταν, ή δεν ήταν επαρκώς όσο θα έπρεπε και αν ήταν πιο συνδεδεμένη με τα αποτελέσματα τότε τα αποτελέσματα θα ήταν καλύτερα εάν λοιπόν έχουμε τώρα τέτοιες πληροφορίες στο χέρι μας είμαστε σε θέση τώρα μέσα στην περίοδο του προγραμματισμού να πούμε ορίστε αυτά είναι τα αδύναμα σημεία τα οποία μπορούν να διορθωθούν μέσα, στην, μέσα σε μια συγκεκριμένη περίοδο χωρίς να περιμένουμε το τέλος της, της περίοδου. Διότι αλλιώς, και ζητώ συγγνώμη, αλλά αυτή η αξιολόγηση είναι πια αυτός δηλαδή δεν προσφέρει τίποτα. Δεύτερο. Χαίρομαι διότι το έγγραφο δείχνει ότι υπάρχουν μέθοδοι διαφορετικές και διαφορετικά φαινόμενα. Οι οικονομολόγοι πάντοτε ε, μαλώνουν για το ποια μέθοδος είναι καλύτερα, καλύτερη. Αλλά αυτό γίνεται χωρίς να ξέρουμε ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα, η χρησιμοποίηση διαφορετικών μεθόδων είναι καλό. Είναι καλή υπόθεση. Αλλά η αξιολόγηση θεωρώ ότι θα δείξει ότι σε ορισμένου τομεί το κριτήριο της ισότητας των φίλων είναι καλό και αλλού δεν έχει επιρροή. Νομίζω ότι αυτό πάλι εδώ το διαβάζει κανείς ανάμεσα στις γραμμές όπως λένε. Και μια τελευταία παρατήρηση. Ή μια ερώτηση προς την Κατερίνα. Γράφεται εδώ στο κείμενο ότι οι περιοχές της υπαίθρου δεν ορίζονται ξεκάθαρα. Αυτά τα λέει η Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο ή η Γενική Διεύθυνση Άγκρι Ή συμφωνούν και οι δύο ότι ο ορισμός δεν είναι ξεκάθαρος. Ο κ. Βλάσεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι είναι σαφές από την παρουσίαση αυτή ότι αν δεν έχουμε όλα τα αποτελέσματα θα είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε ε, συνολικά συμπεράσματα. Ωστόσο, έχω κάποιες ερωτήσεις και ένα σχόλιο για, την, για τον ορισμό των περιοχών της Πέθρου. Πριν από κάποιους μήνες, εδώ στο Κοινοβούλιο είχαμε μία έκθεση για τις αστικές περιοχές και συμφωνήσαμε ότι βάσει των ιστορικών εξελίξεων και των ε, ε, εξελίξεων στα διάφορα κράτη-μέλη θα ήταν δύσκολο να ορίσουμε μια περιοχή και αυτό αποφασίσαμε ότι είναι αρμοδιότητα της κάθε χώρας. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ισχύσει η ίδια προσέγγιση και για τις περιοχές της υπαίθρου. Αυτή θα πρέπει να παραμείνει η αρμοδιότητα λοιπόν των κρατών μελών. Η ερώτηση μου είναι εξή. Έχετε διαπιστώσει προγράμματα εφαρμογής όσον αφορά στην έγκριση, στη χρηματοδότηση και τα θέματα ελέγχου. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και επίσης, έχετε λάβει υπόψη ε, σχόλια των τελικών χρηστών των προγραμμάτων. Η αξιολόγηση εξέτασε καθόλου αυτό το θέμα. Και ε, πότε θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι στις αρχές του επόμενου έτους. Πότε θα είναι διαθέσιμη. Θα έχει κάποια επίπτωση στην τρέχουσα περίοδο. Αυτό το ανέφερε και ο συνάδελφος, ο κύριος Όλμπριχτ. Υπάρχει δυνατότητα να κρίνουμε την αποδοτικότητα των κονδυλίων που δαπανώνται για αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να συγχαρώ τις δύο κυρίες για την ε, πολύ σαφή παρουσίασή τους ε, που ήταν και χωρίς ανοησίες αν μου επιτρέπετε. Στα θεματικά μπλοκ είχατε έξι διαφορετικές ε, τομές, περιοχές Πιστεύετε ότι θα τα σχεδιάσουμε διαφορετικά ω αποτέλεσμα των ερευνών που γίνεται, παραδείγματο χάρη κυρίω για τα περιβαλλοντικά θέματα και την αλλαγή του κλίματο. Δεύτερον, αναφέρθηκε ήδη το θέμα της δυσκολίας του ορισμού των περιοχών της υπαίθρου, αλλά με εξέπλησε το γεγονός ότι ήδη το 25% της χρηματοδότησης πήγαινε στις περιοχές της υπαίθρου. Πιστεύετε ότι θα αυξηθεί αυτό το ποσοστό στα επόμενα χρόνια. Και μια τρίτη ερώτηση Είπατε και παρατήρησαμε πολύ ενδιαφέρον ότι η σύγκριση του κόστους από χώρα σε χώρα ποικίλει. Μήπως μπορείτε να μας πείτε περισσότερα πράγματα για τις διαφορές με καταξατή χωρών μελών. Ποιες είναι οι πιο αποδοτικές από πλευράς κόστους, ποια είναι η πιο ακριβή, ποια είναι η πιο φθηνή. Ο κύριος ε, Βανελίστερ Λόι. Μία επιπλέον ερώτηση. Όταν βλέπει κανείς ότι δεν υπάρχει στρατηγική εστίαση και συγκέντρωση των πόρων με κριτήριο αποτελεσματικότητα, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί πού βρίσκεται το λάθος. Είναι θέμα κανονισμών, είναι θέμα εθνικών προγραμμάτων πλαισίων ή μήπω είναι στο τοπικό επίπεδο το λάθος, στο περιφερειακό. Τι μηχανισμός, εδώ αφού μιλάμε για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, τι είδους μηχανισμός χρειάζεται για να για να υπάρχει περισσότερη εστίαση. Εμείς στο Κοινοβούλιο θέλουμε πάντοτε να έχουμε μια ακριβέστερη, όσο το δυνατόν ακριβέστερη διατύπωση του τι είναι επιλέξιμο και τι όχι. Και στο τέλος καταλήγουμε σε κάτι το άμορφο. Άχαρο πράγμα αυτό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε κάπως πού βρίσκεται το λάθος. Πού είναι η ευθύνη, ε, τοπικό επίπεδο, περιφερειακό, εθνικό, ενωσιακό. Μην ξεχνάτε ότι τα εθνικά στρατηγικά προγράμματα άρχισαν από το 2007 μόλις. Λοιπόν, δεν περιλαμβάνονται δηλαδή στην αξιολόγηση. Δεν έχει κανείς άλλο ζητήσει το λόγο. Κλείνει ο κατάλογος, ναι. Ωραία. Σύνοψη. Θα προσπαθήσω και εγώ να σας τα πω ρητά όπως και εσείς. Λοιπόν, και η Βερονίκη αν χρειαστεί θα συμπληρώσει, αν έχω παραλείψει τίποτα. Είναι το θέμα της κότας και του αυγού εδώ. Βρισκόμαστε στη μέση χρονολογικά, όχι ως προς το προγραμματισμό, στα μέσα της τρέχουσας περίοδου και παρόλα αυτά έχουμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα της εκτονιστέρων αξιολόγησης της προηγούμενης περίοδου. Δυστυχώς έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν έχουμε το καταλληλότερο δυνατό χρονικό πλαίσιο. Δεν θα δοθεί δυνατότητα δηλαδή σε αυτή την περίοδο να διορθωθούν τα λάθη της προηγούμενης. Αλλά μπορούμε ήδη να δούμε, θα μπορέσουμε να δούμε ήδη για την περίοδο 7 με 13 τι θα έπρεπε να αποφευχθεί σε σύγκριση με την προηγούμενη. Επίσης θα προσπαθήσουμε πολύ σοβαρά να έστω και στα μέσα αυτής της τρέχουσας περίοδους να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματά μας τουλάχιστον για τη δέσμη οικονομικής ανάκαμψης έτσι ώστε να δοθεί μια ευκαιρία για κάποια επανεξέταση με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές κάποιας αναπροσαρμογής που ίσως να χρειαστεί. Επίσης τον πρώτο γύρο της καινούργιας διαπραγμάτευσης θα δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε με τις διαχειριστικές αρχές μήπως χρειαστεί αναδιάρθρωση των προτεραιοτήτων. Και εμείς μαθαίνουμε από την αξιολόγηση, ελπίζουμε και οι άλλοι και θα επηρεάσουν τα συμπεράσματα όχι μομεν τις, τα βασικά θεμέλια της πολιτικής αυτής αλλά για, θα επηρεάσουν τα περιθώρια που έχουμε και ίσως διορθωθεί η εστίαση. Και τρίτον, για την επόμενη περίοδο φυσικά θα ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα πλήρως. Όπως είπαμε το Μάρτιο θα γίνει η πλήρης αξιολόγηση, θα ολοκληρωθεί θα γίνει η τελική σύνθεση και τότε με χαρά θα ξανάρθουμε να τα πούμε. και να ακούσουμε τα σχόλιά σας. Οι υπαίθριες περιοχές και οι ορισμοί που τους αφορούν. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες εφαρμόζουν την ε, τρέχουσα ορολογία, αλλά γενικότερα η ακαδημαϊκή κοινότητα δέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα στον ορισμό του τι είναι η υπεθύρια περιοχή. Το είπε και ο κύριος Βλάσανκ. Υπάρχουν και θέματα εθνικών ε, ιδιαιτεροτήτων και ευαισθησιών. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ο καταλληλότερος δυνατός ορισμός όταν η κατάσταση είναι τόσο διαφορετική από χώρα σε χώρα οι εμπειρογνώμονες συνεργάστηκαν με διάφορους ενδιαφερόμενους και αλλά όταν με ρωτάτε ποια ήταν η χρήση των κονδυλίων και ποιο σύστημα ελέγχου εφαρμόστηκε, αυτό δεν αποτελεί τμήμα της αξιολόγησής μας. Μιλάμε μόνο για τα συστήματα εφαρμογής, όχι για την αποτελεσματικότητα ακόμη της χρήσης. Ήταν αξιολόγηση ιδιαίτερα για να μπορέσουν οι καινούργιες χώρες μέλη να εφαρμόσουν αμία αρκετά σωστή δομική αρχιτεκτονική για να χρησιμοποιήσουν, να απορροφήσουν επαρκώς τα κονδύλια. Και αυτό επετεύχθη. Και ένα δεύτερο στόχος ήταν το κανονιστικό πλαίσιο που υπάρχει τι επιπτώσεις, τι αποτέλεσμα έχει, αλλά δεν αφορά αυτό την εκ των υστέρων αξιολόγηση του παρελθόντος. Όσο για το κόστος αναμονάδα δεν έχουμε ακόμη αρκετά στοιχεία για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε ποια μονάδα είναι αποτελεσματικότερη. Γιατί και αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από το γενικότερο πλαίσιο. Κάτι που ισχύει για ένα χρόκτημα με καλαμπόκι μπορεί να μην ισχύει για ένα έδαφος όπου θέλουμε να οικοδομήσουμε μια σύραγγα πούμε. Θα μπορούσε βέβαια να οργανωθεί αλλιώς η τράπεζα δεδομένων για να λαμβάνει υπόψη της και τέτοιες διαφορές αλλά αυτό θα χρειαπετούσε τεράστια επένδυση. Ίσως όμως να φανεί ότι χρειάζεται. Θα το δούμε. Η χρησιμοποίηση του Περιφερειακού Ταμείου στην Ήπεθρο. Ε, γι' αυτό έγινε μια πολύ μικρή μελέτη. είναι βέβαια εδώ η κυρία Ντέλ που έθεσε το ερώτημα, αλλά ήταν πολύ μικρού μεγέθους η μελέτη και δεν σκόπευε να, δει, να αποτιμήσει τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στην ανάπτυξη της υπαίθρου, αλλά απλώς ποια είναι η παρουσία του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου στην Ήπεθρο. Στην τρέχουσα περίοδο παραδείγματο χάρη, που είναι διαφορετική κατάσταση σε σύγκριση με την προηγούμενη, η Γενική Διεύθυνση Γεώρ Άγκρη ε, διαχειρίστηκε ένα αγροτικό ταμείο σε βαθμό πολύ ψηλότερα από το Γενικό Ενωσιακό Περιφερειακό Ταμείο. Άρα δεν εξυλογούμε γενικότερα την αποτελεσματικότητα, αλλά ένα πολύ μικρό δείγμα υποσύνολο. Ίσως η Βερονίκη μπορεί να μας πει τι ακριβώς εύρους ήταν η μελέτη αυτή. ήταν σχεδόν δειγματοληπτική. Δεν είμαι σίγουρος για το ερώτημα του κυρίου Βανίστελ Ρόι, αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι εδώ, οπότε... Α, να προσθέσω εγώ κάτι. Οι διαχειριστικές αρχές έτυχαν διαβούλευσης για την αξιολογική έκθεση, όχι βέβαια ως προς τη διαπραγμάτευση, αλλά τους δόθηκε η έκθεση και η δυνατότητα να τη σχολιάσουν ή να τη διορθώσουν. Τώρα για τις θεματικές ενότητες και την τάξη των προτεραιοτήτων βασίστηκε στην προηγούμενη μεν περίοδο αλλά όντως ε, σε αυτές τις ενότητες δαπανήθηκαν τα περισσότερα χρήματα. Αυτό θελήσαμε να προσέξουμε. Ποιο ήταν το άλλο. Α, ναι. Είναι εκπληκτικό ότι το 25% είναι χαμηλό. Αλλά αυτό γιατί χρησιμοποιήσαμε περιφέρειες που ορίζονται από τον ΟΣΑ ως ύπεθρος. Μπορεί να υπάρχουν περιφέρειες που είναι ύπεθρος αλλά δεν θεωρούνται επίσημα τέτοιες. Όσο για την έλλειψη στρατηγικού εστιασμού, η έκθεση δεν διαπίστωσε ότι υπάρχει τέλεια, τέλεια τέτοια έλλειψη, αλλά ότι δεν είναι ολοκληρωμένη ο εστιασμός. Βέβαια πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η αξιολόγηση αυτή δεν είναι η μόνη που έχει γίνει, δεν είναι το μόνο, η μόνη πηγή πληροφοριών που έχουμε, υπάρχουν κι άλλες. Και τα αποτελέσματά της δεν είναι Ευαγγέλιο, βασίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία και πρέπει να δούμε να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα και με βάση τα στοιχεία που είχαμε για να δούμε τι πρέπει να γίνει. Εμείς πάντοτε με χαρά μπορούμε να πλησιάσουμε εκπροσώπους των χωρών μελών, να συζητήσουμε τις, τα αποτελέσματα μαζί τους. Στην Πολωνία έχει ήδη γίνει αυτό, στην Αυστρία και σχεδιάζουμε και για την Ιταλία ώστε τα αποτελέσματα να χρησιμοποιηθούν από τη συζήτηση που θα γίνει μέσα στα κράτη-μέλη, όχι μόνο στις Βρυξέλλες τέλος. Αν υπάρχει κάποιο λάθος στον προγραμματισμό ή όχι. Βλέποντας τις πρώτες αξιολογήσεις διαπιστώνουμε ότι όταν σχεδιάζεται η στρατηγική, καμιά φορά υπάρχει υπερβολικό εστιασμός στο πού θα δαπανηθούν τα κονδύλια και όχι αρκετά στο τι ακριβώς θα άλλαζε από τι δαπάνες αυτές. Αν γίνει η κατανομή με τον α ή τον β τρόπο. Αυτό πρέπει στο μέλλον να το λάβουμε υπόψη μας, αν είναι δυνατόν. Περισσότερη έμφαση δηλαδή στο τι θα άλλαζε αν δαπανούνταν τα χρήματα όπως έχει προβλεφθεί. Αν αυτό δεν λαμβανόταν υπόψη ήδη από την πρώτη φάση του σχεδιασμού θα ήταν καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ Βερονίκη, δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα άλλο σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους της Κομισιόν και ελπίζω η έκθεση του Μαρτίου να είναι το ίδιο ενδιαφέρουσα Εν τω μεταξύ από ό,τι κατάλαβα οι, περισσο... οι πρόσθετες πληροφορίες θα δίνονται από το ίντερνετ, από την ιστοσελίδα. Ναι, να, εκεί έχει τις διευθύνσεις. Εκεί, ναι. ναι, αν χρειάζεται όμως να τη ζητήσουμε δίνονται και γραπτός. Να, μάλιστα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και καμιά ακρόαση με τους αξιολογητές τους ίδιους. Γιατί με την πολιτική συνοχής μπαίνουμε σε καινούργια νερά. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς πρέπει να γίνει και αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Δημιουργούνται νέα πρότυπα ευρωπαϊκής πολιτικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα οι συντονιστέ